Cominciamo i nostri lavori. Eh, abbiamo qui con λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω τον Υπουργό. Είχα ήδη την ευκαιρία να τον συναντήσω στην Κύπρο πριν δύο μέρες ε, στα πλαίσια της αντιπροσωπείας της ΚΟΖΑΚ. Μπορέσαμε και συναντηθήκαμε και γι' αυτό τον χαιρετίζω για μια ακόμη φορά. Τον καλωσορίζω ανάμεσά μας Καλωσορίζω επίσης και τους υπαλλήλους ε, της Ιταλικής Διοίκησης που μας επισκέπτονται, δημόσιας διοίκησης ενώ. Χωρίς λοιπόν περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Ο κύριος Υπουργός θα μας παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την κατάσταση στα πλαίσια της Προεδρίας του εξαμήνου του θέτοντας ε, τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Μετά την ομιλία του κυρίου Υπουργού, οι συνάδελφοι μπορούν να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Έχετε το λόγο. Dear Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με το σημαντικό έργο το οποίο επίσης φέρει σε πέρας και η Συνταγματική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση και τη θεσμική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται στην αρχή της Κυπριακής Προεδρίας. Πολλοί από εσά γνωρίζουν πόσο προσιλωμένος είμαι στα θέματα της θεσμικής εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Προεδρία είναι μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε μια σημαντική συμβολή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτή την ευκαιρία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας θα λειτουργήσουμε καθαρά ως Προεδρία με θετικό πνεύμα και με στόχο να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα και να αντιμετωπίσουμε το φάσμα αυτό των πολύ σημαντικών θεμάτων που έχουμε ενώπιόν μας, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες απαντήσεις στις πολυμερείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και οι πολίτες της. Σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κέρυας σημασίας. Δεν σημαίνει αυτό ότι η πρόκληση αφορά μόνο την Προεδρία, την Κυπριακή Προεδρία, αφορά όλους μας, ο καθένας στο δικό του τομέα πρέπει να πράξει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Φυσικά, περισσότερο από ποτέ, η Προεδρία χρειάζεται την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε φυσικά να εργαστείτε σε πολλούς τομείς χωρίς την Προεδρία, αλλά η Προεδρία σας χρειάζεται για τις συγκεκριμένες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ένα πνεύμα ευθύνης σε όλους μας και πολλές φορές ακούμε να μας λένε ότι ίσως είναι υπεραισιόδοξη η αντιμετώπιση της Κυπριακής Προεδρίας, γιατί είναι αλήθεια ότι εφορούμαστε από τον ενθουσιασμό μιας χώρας που για πρώτη φορά αναλαμβάνει την Προεδρία. Πιστεύουμε όμως ότι ο ενθουσιασμός μας μπορεί να είναι θετικό και το μήνυμά μα είναι ότι πρέπει να εργαστούμε προ την κατεύθυνση μιας καλύτερης Ευρώπη, μιας καλύτερη Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα γίνει αντιληπτή ως κοντύτερα και πιο ε, σχετική με τους πολίτες της Ευρώπης. Έχουμε αντιμετωπίσει, ιδίως λόγω της χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση μεγάλη ένα μεγάλο αίσθημα ματέωσης και δυσαρέσκειας από τους πολίτες μας, οι οποίοι χρειάζονται τώρα ένα μήνυμα ελπίδας και ιδίως αυτό αφορά τη νέα γενιά στην Ευρώπη. Το γενικό στρατηγικό πλαίσιο της εργασίας μας για μια καλύτερη Ευρώπη θα προωθηθεί μέσω μιας πλειάδας προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, 40 προτεραιοτήτων, οι οποίες έχουν λάβει υπόψη όλα τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο και στο Συμβούλιο, όσο και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα των προσφάτων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Μια πρώτη διάσταση λοιπόν σε αυτές τις προκλήσεις είναι το να έχουμε μια Ευρώπη η οποία θα είναι πιο αποτελεσματική και βιώσιμη. Δεύτερον, θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη η οποία να είναι πιο αποτελεσματική στο οικονομικό επίπεδο, δημιουργώντας απασχόληση και μεγένθηση. Τρίτον, θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη. Μια Ευρώπη η οποία θα είναι πιο κοντά στους πολίτες της, θα έχει αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Τέταρτον, μια Ευρώπη στο παγκόσμιο στερέμα που θα είναι πιο κοντά στους γείτονές της. Αναγνωρίζουμε και έχουμε απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι η επιτυχία της Προεδρίας, όπως είπα και προηγουμένως, συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα και την ένταση της συνεργασίας που θα πρέπει να έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θεσμικό σας όργανο εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και παίζει ένα ζωτικό ρόλο για την επίτευξη οποιοδήποτε, για την επιτυχία οποιοδήποτε εγχειρήματο το οποίο τυχόν να αναλάβουμε. Έχουμε ξεκινήσει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε πολλές επαφές και στην Κύπρο και εδώ στις Βρυξέλλες και είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία αυτή ενισχύει πράγματι τις σχέσεις μας και βασίζομαι σημαντικά στη σημερινή μας συνάντηση για να συνεχίσουμε αυτήν την θετική και παραγωγική σχέση. Έχουμε λοιπόν δεσμευτεί για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος και ο συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υποστηρίζουμε τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως απορρέει από τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι πάντα πληροφορημένο και θα μπορεί να συμμετέχει ήδη σε πρώιμο στάδιο σε όλα τα εγχειρήματα. Έχουμε κάθε σεβασμό για την ενωσιακή μέθοδο, για το ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πάντα κινούμεθα μέσα στο πνεύμα των συνθήκων. Πιστεύω ότι αυτός είναι και ο βέλτιστος τρόπος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ως Προεδρία αποδίδουμε τη μεγαλύτερη σημασία στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παίρνουμε πολύ στα σοβαρά το ρόλο που επομιζόμεθα ως Προεδρία. Έρχομαι τώρα στα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες της Συνταγματικής Επιτροπής. Καταρχήν θέλω να χαιρετήσω την έναρξη της διαδικασίας της ε, πρωτοβουλίας πολιτών από τον Απρίλιο του ενεστώτος έτους και θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν για την πρόοδο που επέτυχε. Όλα αυτά φέρνουν την ε, Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και επιτρέπουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους και το αίσθημα ότι συμμετέχουν και αυτοί στα τεκτενόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι η καλύτερη εγγύηση για τη συνέχιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Θέλω επίσης να συγχαρώ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τη συμφωνία που επιτεύχθη κατά την Δανική Προεδρία για την διαθεσμική συμφωνία που εμπλέκει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την πρόσβαση <clears throat> από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε διαβαθμισμένα έγγραφα σε θέματα άλλα από αυτά που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Η προετοιμασία για την εφαρμογή αυτού του μέτρου συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές και στα δύο όργανα. Υπάρχει από ό,τι γνωρίζω η έκθεση του κυρίου Χάφνερ, η οποία θα ψηφιστεί σήμερα για το θέμα αυτό. Η συνεργασία σε τεχνικό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υποφέλης και πιστεύουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του ενεστώτος έτους θα περατωθεί αυτή η διαδικασία και η συνεργασία των δύο οργάνων θα αρχίσει εγκαίρως. Όπως γνωρίζετε επίσης, ένα κέριο στοιχείο της διαθεσμικής αυτής συμφωνίας που συνήφθη τον Φεβρουάριο είναι και η δέσμευση του Συμβουλίου ότι θα αποδεχτούμε <clears throat> και θα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση της διαθεσμικής συμφωνίας του 2000 μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου σε σχέση με την πρόσβαση από το Κοινοβούλιο σε ευαίσθητα θέματα ε, που αφορούν την πολιτική άμυνας και ασφάλειας ως Προεδρία εμείς θα τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και να προωθήσουμε τις σχετικές συζητήσεις με πλήρη σεβασμό του ρόλου της ΙΠΑ ε, της εκπροσώπου και αντιπροέδρου κυρίας Άστον σε ό,τι αφορά τα θέματα της ΚΕΠΑ. Σήμερα βέβαια είναι και μια ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με θέματα που βρίσκονται στο κοινό μας θεματολόγιο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Και θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, να εστιάσω στα εξή σημαντικά θέματα. <clears throat> τα δικαιώματα έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και η προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή ε, Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μάρτιν, δεν ξέρω αν είναι παρόν εδώ σήμερα, και τα άλλα μέλη της ε, ομάδος διαπραγμάτευσης, ιδίως τον κύριο Νταφ και τον κύριο Βίλαντ, για, τις πάρα πολύ, για την πάρα πολύ επικοδομητική συνάντηση που είχαμε χθε. Με τη συζήτηση αυτή είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε ε, τα θέματα που μας ενδιέφεραν και να δούμε τον δρόμο προς τα εμπρός. Είμαστε απόλυτα προσφυλωμένοι να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέραση η Ιδανική Προεδρία για τα θέματα αυτά και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές απόψεις και ότι είναι δύσκολα και ευαίσθητα τα θέματα αυτά. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και την διαπραγματευτική ομάδα για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τα, τις διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των οργάνων μας, των θεσμικών μας οργάνων, με στόχο να πετύχουμε εγκαίρως μια λύση για τα θέματα αυτά. Θα πράξουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν για να καταλήξουμε σε ένα αίσιο πέρα σε αυτή τη διαδικασία, όπως ανέφερα και χθε. <clears throat> Πιστεύουμε το δικαίωμα έρευνας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα σημαντικό στοιχείο των εποπτικών εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμβάλλει στην περαιτέρω προώθηση των αρχών της λογοδοσίας και της διαφάνειας. Σεβόμαστε πλήρως το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να έχει εξεταστικές επιτροπές στις οποίες θεσμεύει και επίσης το να ε, θεσπίζει τις εξειδικευμένες ρήτρε που διέπουν αυτές τις επιτροπές. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει και από τις ε, συνθήκες. Πιστεύουμε ότι μπορούμε μέσα στα πλαίσια των συνδικών να βρούμε μια λύση για όλα αυτά τα θέματα και να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα είναι αμοιβαία αποδεκτή, αποδεκτή και από τα τρία μεγάλα θεσμικά όργανα. Μέσα στο πνεύμα αυτό λοιπόν είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα πάντα μέσα στο πνεύμα αυτό του ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο τους πολίτες της, που είναι και ένα από τα κύρια μηνύματα της Κυπριακής Προεδρίας, είναι πεποίθησή μας ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι η διαμόρφωση και η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και η επίτευξη της έκφρασης της, ε, των απόψεων των πολιτών είναι κάτι το οποίο είναι ένας βασικός στόχος της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει πρόθεση να προτείνει ένα νομοθετικό πακέτο που θα περιλαμβάνει ένα κανονισμό ο οποίο δίδει νομική προσωπικότητα στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και επίσης τροποποίηση υφισταμένων κανονισμών σε σχέση με τους κανόνες που διέπουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εγκαίρως όλοι αυτοί οι κανόνες πριν από τις ευρωεκλογέ του 2014. Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπεται για το Σεπτέμβριο του ενεστώτος έτους. Το Συμβουλίο θα εξετάσει προσεκτικά την πρόταση αυτή μόλις διατυπωθεί και διαβιβαστεί στο ενδιάμεσο διάστημα εμείς συνεχίζουμε τις επαφές μας με την Κομισιόν σε σχέση με το χρόνο-διάγραμμα και ορισμένες πτυχές αυτής της πρότασης και είμαστε όπως είπα απόλυτα προσιλωμένοι στο να συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να υπάρξει η έγκριση αυτής της νομοθετικής πρότασης εγκαίρως πριν από τις ευρωεκλογέ και είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να τηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει επίσης το θέμα της πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο προκύπτει από το άρθρο 6 της ε, Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το θεωρούμε μεγάλο επίτευγμα της Συνθήκης της Λισαβόνας. Για πρώτη φορά στην ιστορία όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υφίστανται την ίδια εξέταση όπως και αυτά τα οποία λαμβάνουν 47 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων και όλα τα κράτη-μέλη. Για πρώτη φορά κάθε Ευρωπαίος πολίτος μπορεί να προσφύγει κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Αυτό θα προστατεύσει βέβαια τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο. Τονίζει την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωση για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και επίσης ενισχύει τον ρόλο μα ως ε, ενός ε, προσιλωμένου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεωρώ πως σύμφωνοι πλήρως επίσης με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και τι εννοώ, να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Όσον αφορά λοιπόν την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, ε, ΕΣΔΑ, χρειαζόμαστε ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και την, συμφωνή, και την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως των Εθνικών Κοινοβουλίων. Καλωσορίζουμε τις ε, πρόσφατες λοιπόν εξελίξεις προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ η αρμόδια ομάδα εργασία του Συμβουλίου συνεχίζει τη συζήτηση επί των αρχών που θα κατευθύνουν την Κομισιόν όταν θα παρουσιάσει την πρότασή της για τους εσωτερικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ρυθμίσουν την συμπεριφορά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του ΕΔΑΔ. Ευχαριστούμε λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι εκφράζει την στήριξή του για την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τον Μάιο του 2010, η οποία επαναλήφθηκε τον Απρίλιο του 2012. Είμαστε πεπισμένοι πως ε, όταν εργαζόμαστε μπορούμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και η Προεδρία της Κύπρου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διευκολύνει αυτή την συμφωνία. Αυτό σημαίνει βεβαίως πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται πάντα ε, εγκαίρως για την πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων. Να επαναλάβω πως ε, θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την συνεργασία μας και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εργαστούμε για μια καλύτερη Ευρώπη και γνωρίζω επίσης πως έχετε και άλλα θέματα να ασχοληθείτε. Και παραμένω στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε οτιδήποτε ε, σημαντικό αυτή τη στιγμή. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους οι οποίοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά στο τέλος μπορείτε να δώσετε μια συνολική απάντηση. Κύριο Σταρκόσκη έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ειλικρίνειά σας και τις ε, παρατηρήσεις σας βασιζόμαστε στην ε, Κυπριακή Προεδρία, ειδικά για τα θέματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Αναφερθήκατε σε περισσότερα από αυτά στις διερευνητικές επιτροπές. Ξέρετε πως είχαμε κάποια προβληματάκια και ελπίζουμε η Κυπριακή Προεδρία να δεχτεί τα επιχειρήματά μας και βεβαίως ε, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Η άποψή μας είναι πως θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και καμιά φορά έχουμε την αίσθηση πως το Συμβούλιο επιλέγει να διατηρήσει το status quo, το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό. Για τα πολιτικά κόμματα θα θέλουμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με τρόπο καινοτόμο. Θέλουμε να μπορούν να φαίνονται επιτέλους τα πολιτικά κόμματα και, γιατί... και θέλουμε οι ευρωεκλογέ βεβαίω να έχουν θέμα τα ευρωπαϊκά θέματα υπό την αιγίδα των πολιτικών κομμάτων μας για να αρχίσουν να μπαίνουν ευρωπαϊκά θέματα στην συζήτηση. Αυτή είναι μια προτεραιότητά μας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω για αυτά τα οποία δεν αναφέρατε και τα οποία οπωσδήποτε μας απασχολούν ε, για την αρχιτεκτονική δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, για το έγγραφο Φαν και τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προετοιμάζουμε εκθέσεις για την οικονομική διακυβέρνηση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ε, γι' αυτό είμαι υπεύθυνο εγώ και ο κύριος Γκουαλτιέρη σε αυτή την επιτροπή και θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώς βλέπετε τη δική σας εμπλοκή ως ε, Προεδρία της Κύπρου στις συζητήσεις αυτές και ποιες είναι οι προτεραιότητε σας όταν ε, μιλάμε για την αρχιτεκτονική η οποία θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας, δηλαδή αν μπορούσατε να πείτε ποιους κανόνες ε, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε στην όλη διαδικασία, πώς θα ορίζατε εσείς την επιτυχία σας όσον αφορά το να επηρεάσετε τη συζήτηση, κάτι το οποίο βεβαίως δεν θα είναι εύκολο για την Προεδρία για λόγους ε, προφανείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριος Γκουερέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για την έλευσή σας ενώπιον της Επιτροπής μας για να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι θέσεις σας και ποιες είναι οι προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, εμψυχώσω, να σας παροτρύνω στη συνέχιση των προσπαθειών σας σε αυτή την πρώτη προεδρία της χώρας σας. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό με τον οποίο ξεκινάει πάντα μια χώρα την πρώτη της Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω και προσωπικές αναμνήσεις από την εποχή που για πρώτη φορά ανέλαβε το 1989 την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ισπανία τότε ήμουνα επικεφαλής του γραφείου του Υπουργού Παιδείας της Ισπανίας, ο οποίος στη συνέχεια έγινε ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Σολάνα. Θυμάμαι πολύ καλά το πώς είχε συμμετέσχει όλη η χώρα, όλη η κοινωνία, είχε κατεβάλει προσπάθειες για μια επιτυχή προεδρία. Επομένως ήταν μια πραγματική ε, πρόκληση για όλους και φυσικά εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα ότι είσαστε μια σύντομη προεδρία γιατί είσαστε στο δεύτερο εξάμεινο του έτους. Σε σχέση με αυτά που ανέφερε και ο κύριος ε, Ταρκόφσκι, η παρέμβαση του Προέδρου του, Ευρωπαϊκού, του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28 ε, και 29 Ιουνίου ήταν μια ακόμα υπόμνηση και υπογράμμιση του γεγονότος ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια διαδικασία βαθιάς θεσμικής μεταρρύθμισης των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός προβληματισμού για αυτή τη μεταρρύθμιση, όπου συμμετέχει ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο πρόεδρος της Ευρωομάδος του. Αλλά όπου ελείπει οποιαδήποτε πραγματική παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η θέση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ότι Ακριβώς όταν εμπλεκόμεθα σε μια διαδικασία η οποία πρέπει να οδηγήσει σε μια πολιτική ένωση, μια πολιτική ένωση η οποία πρέπει να βασίζεται στη δημοκρατική νομιμοποίηση η οποία προκύπτει από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία <clears throat> ενσαρκώνεται, αν θέλετε, με άμεσο τρόπο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει κάτω από τετοιες συνθήκε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή η οποία εκείνη τώρα και θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω την αίτησή μας ότι από την πλευρά της Κυπριακής Προεδρίας θα πρέπει να υπάρξει μια, ένα θετικό κλίμα για μια μεγαλύτερη συμμετοχή και παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπατε και στα εισαγωγικά σας σχόλια. Σε ό,τι αφορά τώρα στην πρόσβαση, στην προσχώρηση καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, αυτή είναι μια διαδικασία στην οποία εγώ είμαι ο αρμόδιος από την Επιτροπή μας, ο οποίος παρακολουθεί τη διαδικασία διαπραγματεύσεων που ασκεί η Κομισιόν. Θα ήθελα να τονίσω ότι φαινόταν να έχουμε πριν από μερικούς μήνες ήδη επιτύχει μια συμφωνία. Αλλά κάπως αδρανοποιήθηκε αυτή η συμφωνία στο Συμβούλιο λόγω της αντίδρασης ορισμένων κρατών μελών Φαίνεται ότι τώρα διαφαίνεται και πάλι η δυνατότητα να προχωρήσουμε και η Κομισιόν έχει επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Συμβουλίο της Ευρώπης. Θα ήθελα λοιπόν και στο θέμα αυτό να σας ζητήσω να συνεχίσετε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ιδανική Προεδρία προς την κατεύθυνση αυτή και να προσπαθήσετε να πείσετε τις χώρες ακόμα αυτές που εξακολουθούν να έχουν δισταγμούς μέσα στο Συμβούλιο ότι πρέπει να περατωθεί αυτή η διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο της Ευρώπης εμείς από την πλευρά της ε, Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα να μπορέσει να περατωθεί η διαπραγμάτευση αυτή πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην χρειαστεί μετά από το 2014 να εμπλακούμε και πάλι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης τη στιγμή που ήδη κρατάει δύο, μισή χρόνια σχεδόν η διαπραγμάτευση. Ξέρω τώρα ότι η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι πάντα εύκολη. Θα θέλαμε όμως να σας ζητήσουμε να βοηθήσετε όσο μπορείτε να υποστηρίξετε τις, ε, τα αιτήματα, τις ε, εκκλήσεις που έχει διατυπώσει η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2013. Οι αιτήσει μας συνάπτονται περισσότερο με τα θέματα επικοινωνίας προς τους πολίτες με την ε, διαμόρφωση ενός συστήματος ακροάσεων για τις πρωτοβουλίες πολιτών και για την εκλογική διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί το 2014. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι καλή τύχη. Χαίρομαι που σας συναντώ και εξ ονόματος της ομάδας των φιλελευθέρων κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια και στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου, για τον τριμερή διάλογο, μπορεί να υπάρξει πρόοδος πράγματι. Συμφωνώ με την σημασία την οποία δίδεται στην ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Το θέμα των εσωτερικών κανόνων. Αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος. Νομίζω ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να σημειώσουν κάποια πρόοδο εκεί. γιατί αλλιώς οι διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης μπορεί να καταρρεύσουν. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι τακτικές ρυθμίσεις, θα έλεγα, ενισχυμένη πλειοψηφία, να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή να αντιπροσωπεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Υπουργών Αυτά όλα πρέπει να θεωρηθούν δεδομένα ότι θα συνεχιστεί η ισχύ τους. Είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε τη λογική της συνθήκης της Λισαβόνας. Και γι' αυτό παρακαλώ σαν Προεδρία να είστε όσο σκληροί χρειάζεται και απέναντι στην Βρετανική κυβέρνηση, η οποία δεν φαίνεται να εκτιμά δεόντως το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Είστε ιδιαίτερο ευγενείς απέναντι στην Προεδρία της Δανίας, αναμενόμενο από πλευρά σας. Είναι όμως σαφές ότι τα μπέρδεψαν τα πράγματα σε σχέση με τη νομική βάση για τους εφαρμοστικούς κανονισμούς του Σέγγεν. Μπορείτε παρακαλώ να μας διαβεβαιώσετε ότι θα κάνετε κάθε προσπάθεια από πλευρά σας για να αποκαταστήσετε το status quo που ίσχυε πριν από, την, το λάθος το οποίο διέπραξε η Προεδρία της Δανίας που είναι μια προσβολή εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπονομεύει την ίδια την διαδικασία Σέγγεν. πρέπει να είναι μεγάλη προσπάθεια της Προεδρίας να διατηρήσει την συνεκτικότητα και την πειθαρχία στα εσωτερικά του, στο εσωτερικό του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που ακολουθεί μια συνάντηση κορυφής και στα πλαίσια της οποίας στην ουσία οι Υπουργοί τι κάνουν, συναντιόνται και αρχίζουν και διαλύουν τις αποφάσεις και τις συνενέσεις τις οποίες πιστεύαμε ότι είχαμε καταλήξει κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής. Και αυτό γιατί υποτίθεται δεν είχαν καταλάβει ακριβώς πάνω σε τι είχαν συμφωνήσει. Και αυτό δυστυχώς διότι οι υπουργοί πολλές φορές δεν λειτουργούν με την υπευθυνότητα την οποία αναμένει κανείς από πλευράς τους. Είδαμε πρόσφατα παραδείγματα και από πλευράς των Φιλανδών και των Ολλανδών μετά από τη συνάντηση κορυφής πριν 15 μέρες. Νομίζω λοιπόν ότι σαν προεδρεύοντες θα μπορέσετε να αγριέψετε λίγο. απέναντι στους υπολείπους γιατί πλησιάζουμε σε ιστορικά σημαντικές συναντήσεις του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ένα επιπλέον θέμα στο οποίο δεν αναφερθήκατε και το οποίο είναι δύσκολο να αναφέρει βέβαια κανείς, το δέχομαι, ακόμα και στην Επιτροπή μας. Το θέμα του αριθμού των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα έλθουν από την Κροατία. Θα είναι 11. Αυτή είναι η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε αυτή την περίπτωση από πού θα πάρουμε τα 11 αυτά μέλη. Από πού θα τα βγάλουμε δηλαδή. Ερωτήσεις, ερωτήσεις που ασχολούνται με την ουσία των προβλημάτων. Ευχαριστώ τον κύριο Νταφ. Είναι γνωστός για τον φιλοευρωπαϊσμό του ο κύριος Νταφ παρά την αντίθεση της χώρας του μερικέ φορές προωθεί την ευρωπαϊκή ιδέα. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Έπνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Μαυρογιάννη στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και για τις εξηγήσεις σας για τα της Κυπριακής Προεδρίας. Θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία αναφέρατε και μετά σε ένα το οποίο δεν αναφέρατε όσον αφορά το δικαίωμα έρευνων. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια λύση λογική. Δεν είναι λογικό να έχουμε διερευνητικές επιτροπές εάν το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να διαλέξει και να ακούσει τους μάρτυρες που κρίνει αναγκαίο. Εάν δεν υπάρχουν δυνατότητες για κυρώσεις, εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα και στις απαραίτητες πληροφορίες και είμαι σίγουρος πως υπάρχουν ρεαλιστικές λύσεις για όλα αυτά τα ζητήματα εάν ε, υπάρχει θέληση να καταλήξουμε σε μια καλή θετική λύση. Οπότε βασιζόμαστε στην ε, Προεδρία σας για αυτό το θέμα. Όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τον δημοσιονομικό κανονισμό, νομίζω πως είναι σημαντικό να γίνει αυτό και ταυτόχρονα να κάνουμε ένα βήμα προς πιο δημοκρατικές λύσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο και εντός των κομμάτων. Και θα ήθελα να πω κάποια λόγια για αυτό το οποίο είπατε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, γιατί δεν ξέρω εάν γνωρίζετε ακριβώς τα πράγματα. Η τέθη ενισχύει την 1η Απριλίου, αλλά ακόμα δεν λειτουργεί λαμβάνουμε πολλά παράπονα από ευρωπαϊκές ε, πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν ήδη καταγραφεί έχουν καταγραφεί από την Κομισιόν και δεν μπορούν να μαζέψουν τις υπογραφές. Έχουν ένα περιθώριο 12 μηνών, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν γιατί το σύστημα ακόμα δεν λειτουργεί. Κάποιες πλευρές του υπάρχουν προβλήματα και με το site υπάρχουν προβλήματα με την φιλοξενία ε, στους σερβερ που πρέπει να είναι επιστοποιημένοι. Μετά ε, βεβαίω αυτό είναι κάτι τόσο ακριβό που δεν μπορούν οι πολίτες να το πληρώσουν. Δηλαδή εμείς σκοπεύαμε η πρωτοβουλία αυτή των πολιτών να είναι δωρεάν. Εμείς, εγώ Είμαι σε συνεχή και άμεση επαφή με την Κομισιόν για να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά νομίζω πως μία όθηση από το Συμβούλιο θα βοηθούσε, γιατί ήταν το μεγάλο επίτευγμα της συνθήκης της Λισαβόνας. Είπαμε στο λαό πως θα έχουμε περισσότερη δημοκρατία, εσείς μπορείτε να έχετε πρωτοβουλίες πολιτών και εάν δεν λειτουργήσει αυτό θα έχουμε μεγαλύτερη απογοήτευση παρά ε, εμπλοκή του κόσμου με την Ευρώπη και είναι ωραία πράγματα. Νέοι άνθρωποι που έχουν ε, και έτσι, πιο ιδεαλιστικές ε, αλλά και πολύ ρεαλιστικές προτάσεις και τώρα εκνευρίζονται γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα. Οπότε πιέζουμε και εμείς, αν πιέσετε και εσείς ελπίζω να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Και τέλος, το τελευταίο ζήτημα το οποίο ήθελα να θίξω είναι κάτι το πιο γενικό. Αφορά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα στην Ευρώπη και το μέλλον της Ευρώπης. Και θα έλεγα πως ένα θέμα είναι τα μέτρα διάσωσης, τα έκτακτα μέτρα, τα οποία λαμβάνουμε εδώ και χρόνια, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε πού στοχεύουν όλα αυτά οι πολίτες θα μας ακολουθήσουν μόνο εάν αντιλαμβάνονται ποιος είναι ο στόχος που οδηγούν όλα αυτά. Και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια εικόνα της μελλοντική αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, όπου όλα αυτά θα βασίζονται σε δημοκρατική νόμιμοποίηση. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως είναι δική τους η Ευρώπη, όχι μόνο των θεσμικών οργάνων. Οπότε πρέπει να βρεθεί μια νέα αρχιτεκτονική εντός της κοινοτικής μεθόδου και επί τη βάση της νομοποίησης που παρέχουν οι πολίτες μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον σκοπό αυτό οπωσδήποτε χρειάζεται μια σοβαρή συζήτηση, οπωσδήποτε χρειάζεται μια συνέλευση αλλά όχι μια συνέλευση η οποία θα υπάρχει μόνο για να δεχτεί προτάσεις οι οποίες θα έχουν ήδη ε, καθοριστεί από τους Προέδρους. Χρειάζεται συζήτηση, εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης θα έλεγα πως χρειάζεται να εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία η οποία θα μπορεί να αντλήσει νομιμοποίηση και να προσφέρει δημοκρατία, αν θέλετε, στο πλαίσιο της Ευρώπης. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις, ε, τις επιλογές, το, το προς τα που θα στραφούμε για το μέλλον του της Ευρώπης για τη μελλοντική αυτή αρχιτεκτονική και απευθύνω έκκληση σε εσά και βασίζομαι σε εσά να βοηθήσετε την Ευρώπη να βρεθεί σε ένα καλό δρόμο όπου οι πολίτες ε, θα αισθάνονται μέρος και κυρίαρχοι της Ευρώπης. Σύμφωνα λοιπόν με τη μέθοδο που θα διαλέξετε για τις συζητήσεις αυτές για το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ. Δύο ακόμα ομιλητές έχουμε. Ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν περιοριστήκατε σε θέματα της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, ούτε και εγώ θα περιοριστώ σε αυτά. Είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι κοντύτερα στους γείτονές της. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γείτονες να σταματήσουν να είναι χώρες διέλευσης για παράνομους μετανάστες. Στην περίπτωση της Τουρκίας αυτό μπορεί να είναι δύσκολο από ό,τι καταλαβαίνω και ελπίζω να μην σας ενοχλεί αυτό, η Τουρκία αρνείται να αναγνωρίσει την Προεδρία σας. Εγώ δεν είμαι ακριβώς ο πιο ενθουσιώδης ευρωπαϊστής, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μια απαράδεκτη και ε, μια απαράδεκτη προσβολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η στάση της Τουρκίας. Πέραν αυτού γνωρίζουμε ότι το 1 τρίτο της χώρας σας είναι υποκατοχή. Υπήρξαν ε, καταστροφές και ε, συλλήσεις εκκλησιών στην Βόρεια Κύπρο. Δεν μπορεί λοιπόν η Τουρκία να συνεχίζει να είναι μια υποψήφια χώρα όσο συνεχίζεται η κατοχή της Βόρειας Κύπρου. Είπατε ότι θέλετε να ενθαρρύνετε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και συνειδητοποίηση και να υπάρξει η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα χωριστή από την ευρωπαϊκή ηθαγένεια αλλά πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι μονάχα σαν μια προσθήκη και δευτερεύουσα πέραν της εθνικής συνειδητοποίησης και εθνικής ταυτότητας. Δεν ξέρω όμως πώς θα μπορέσει να ενισχυθεί αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα εάν γίνει μέρος Ευρώπης η Τουρκία η οποία δεν είναι ευρωπαϊκή σε πολιτιστικό ή ιστορικό ε, επίπεδο ούτε καν και γεωγραφικά γιατί 90% του εδάφους της είναι εκτός της Ευρώπης. Αναφερθήκατε στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Κάποια πράγματα που στην αρχή απλώ επιτρέπονται γίνονται σιγά σιγά υποχρεωτικά. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι καταρχήν ότι τα πολιτικά κόμματα θα επιτραπεί καταρχήν η λειτουργία του και μετά θα γίνουν υποχρεωτικά για τι ευρωπαϊκέ εκλογικέ περιφέρειες, για τι ευρωεκλογέ, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σε ευρωπαϊκέ εκλογικέ περιφέρειες και αναρωτιέμαι πόσο θα χρειαστεί μέχρι ότου τα ευρωπαϊκά κόμματα θα είναι ο υποχρεωτικό διάβλο για όσου εκλέγονται στι ευρωεκλογέ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο και φυσικά αυτό δεν <clears throat> προβλέπεται ακόμα, αυτό θα περιορίσει τη δυνατότητα του εκλέγεστε και επομένω εισόδου στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο μόνο σε αυτούς που έχουν μια ευρωπαϊκή στάση και προοπτική. Ακούσαμε και χθε και σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποφασίζει τα θέματα για τα οποία γίνεται η διεκδίκηση της εκλογής της ευρωεκλογές. Τότε τα, ευρωπαϊκού χαρακτήρα κόμματα θα είναι και ο διάβλος μέσα από τον οποίο λαμβάνονται αποφάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα θέματα. Κύριος Μέσα Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαυρογιάννη, καλώς ήλθατε. Εγώ αντίθετα με τον κύριο Νταφ δεν ε, έχω ανάγκη να είμαι ευγενής προς την Δανική Προεδρία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να μας ε, επιβεβαιώσετε ότι η συμφωνία για το καθεστώς του Σέγγερ που ανέφερε ο κύριος Νταφ δεν ήταν μια δανεική απόφαση, αλλά μια ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Τώρα θέλω να θέσω και ένα ερώτημα και αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την παρουσίαση του προγράμματός σας προς την Θεσμική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω ένα ερώτημα σε σχέση με κάτι το οποίο μπορεί να είναι το πιο σημαντικό συνταγματικό θέμα καθ' όλη τη διάρκεια τη Προεδρία σας συγκεκριμένα το να φύγει μια χώρα από την Ευρωζώνη. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό άμα δείτε τον οικονομικό τύπο και αυτά τα οποία είναι οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια, οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην Ευρωζώνη. Οι σημερινές δομές της συνθήκης από τεχνική άποψη δεν επιτρέπουν σε μια χώρα να φύγει από τη ζώνη του ευρώ χωρίς να φύγει από τη σύνολη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της Ελλάδος, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί και από συνταγματική έποψη. Πώς λοιπόν <clears throat> θα το αντιμετωπίσετε αν ανακύψει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Τι είδους προστατευτικά μέτρα μπορείτε να λάβετε ήδη από τώρα, ώστε να αντιμετωπίσετε αυτό το ενδεχόμενα ανακύπτων συνταγματικό θέμα. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα μέσα στην ε, δική σας Προεδρία, θα γίνει μάλλον στην επόμενη Προεδρία και αυτό είναι και προς το καλό της Ελλάδος πιστεύω. Τι προετοιμασίες λοιπόν θα αναλάβετε ώστε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση όταν προκύψει που πιστεύω ότι αναμφίβολα θα γίνει πραγματικότητα σύντομα. Δεν έχω ζητήσει άλλη το λόγο. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Υπουργό, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις να υπογρομίσω κάτι σχετικά με τη γειτονία. και με τις χώρες αναφέρομαι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος βρίσκεται σε μια γεωγραφική κατάσταση θα έλεγα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Βρίσκεται ακριβώς στη γωνία της Μεσογειακής Λεκάνης η οποία είναι αιστεία θα έλεγα ανάφλεξης για πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν τα προβλήματα με τη Συρία, με την Τουρκία, με το Ισραήλ Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσα σε έξι μήνες να μπορέσει κανείς να διορθώσει τα στραβά του κόσμου. Αλλά παρόλα αυτά ίσως να μας πείτε λίγα λόγια για τον ρόλο τον οποίο έχει η Κύπρος, όχι μόνο σχετικά με το συγκεκριμένο εξάμεινο, αλλά και κάπως πιο μακροπρόθεσμα, ιδιαίτερα για την περιοχή σας, ε, από όπου προήλθε θα έλεγα και η Ευρώπη και ρόλος της Ευρώπης δεν είναι μόνο να διατηρεί την ειρήνη στο εσωτερικό της αλλά και να την επιβάλλει αν γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, περισσότερες από τις ερωτήσεις είναι δύσκολες, αλλά αν μου επιτρέπετε, να προσπαθήσω να είμαι όσο δυνατόν πιο ειλικρινής. Οπότε, μην θεωρήσετε πως αυτά τα οποία θα σας πω είναι και 100% η γραμμή του Συμβουλίου. Και ελπίζω η γραμματεία του Συμβουλίου να με συγχωρέσει εάν κάποια στιγμή ξεπεράσω τη γραμμή του Συμβουλίου. Αλλά πρέπει νομίζω να είμαστε ειλικρινεί ε, στις ε, επαφές μας. Και αυτό προσπαθήσω να κάνω σήμερα. Θεωρώ πως όσον αφορά τις διερευνητικές ε, επιτροπές τις εξεταστικές επιτροπές ε, η χθεσινή συνάντηση έδειξε πως μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα και αυτό το ανέφεραν και άλλοι αργότερα, αλλά συμφωνήσαμε πράγματι πως πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο θα είναι αποτελεσματικό, συνεπές και δεν πρέπει να ξεχνάμε το στόχο μας. Στην τελική ανάλυση δεν μπορούμε να έχουμε μια εξεταστική επιτροπή που μόνο στα λόγια πρέπει να βοηθάει τον στόχο της διαφάνειας, ε, τη λογοδοσία, να καταπολεμήσει την ατιμορρησία. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα λοιπόν, αλλά νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε τους ερχόμενους μήνες να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να προχωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη και τις πολιτικές περιπλοκές και τις διοικητικές καμία φορά το καθεστώς των διαφόρων εμπλεκομένων ε, αξιωματούχων της Κομισιόν των κρατών μελών πώς θα υπάρχει σύνδεση μεταξύ εθνικού επίπεδου και του υφισταμένου καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Υπαλλήλου, του Ευρωπαίου Υπαλλήλου. Αλλά σε τελική ανάλυση έχετε δίκιο. Πρέπει να έχουμε κάτι το οποίο θα έχει ουσία. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι απλά για να λέμε ότι το κάναμε. Και ήδη αναφέρθηκε και από τον κύριο Νταφ Ξέρετε πως θεωρώ πως και ο ίδιος ε, μετά τη χτεσινή μας συνάντηση πιστεύει πως ε, είμαστε σε καλό δρόμο για να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα και πραγματικά θα καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Και δεκτώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σχέφνερ για κάτι το ρεαλιστικό αυτό θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Για τα πολιτικά κόμματα. Ξέρετε, θεωρούμε πως υπάρχει κάποια προσθεμένη αξία στο να έχουμε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα, κύριε Μπρόνς, σας διαβεβαιώ πως ε, το σκεπτικό μας δεν είναι να είμαστε τόσο περιοριστικοί. Το θέμα είναι να έχουμε μια προστιθέμενη αξία. Όχι να περιορίσουμε την ε, συζήτηση ή την πρόσβαση στις ε, ευρωεκλογέ ή τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα με το να έχουμε μια ομπρέλα η οποία δεν θα επιτρέπει ακόμα και σε κόμματα τα οποία δεν θα είναι φιλοευρωπαϊκά στόχος είναι να αυξηθεί ο χώρος ελευθερίας ε, στην Ευρώπη. Όλοι είμαστε κατά του, του αντίθετου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και αυτό το οποίο είπατε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και θεωρώ πως για το προσεχές μέλλον δεν υπάρχει ζήτημα του να επιλέξουμε μεταξύ των δύο αυτών. Αυτά τα πράγματα πάνε μαζί για το προσεχές μέλλον. Τώρα εάν η τα πράγματα εξελιχθούν κατά τρόπον ώστε τελικά να έχουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα πάνω από την εθνική ταυτότητα, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω πως αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, βεβαίω εκτιμούν και έχουν και τις δύο ταυτότητες και δεν μπορούμε να καταργήσουμε την εθνική ταυτότητα επειδή προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια ευρωπαϊκή. Κατόπιν, το σημαντικότερο ζήτημα, θεμελιώδες, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους ερχόμενους μήνες, δεν είναι οπωσδήποτε ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Προεδρία. Η Προεδρία έχει το ρόλο της να παίξει, αλλά το ζήτημα αυτό πάει ακόμα παραπέρα. Το θέμα είναι πώς διαμορφώνουμε το μέλλον της Ευρώπης ε, και τη μελλοντική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωση. Και η συζήτηση ξεκίνησε όλοι συνειδητοποιήσαμε πως παραδείγματο χάρη μέχρι το τέλος του περασμένου έτους ε, είχαμε εστιαστεί στην εξυγένση των δημοσίων οικονομικών σε ζητήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας επιτήρησης ε, και μετά ε, αντιληφθήκαμε πως πρέπει να ε, εστιαστούμε στην ανάπτυξη και τις δουλειές και μετά υπάρχει βεβαίως και το δημοσιονομικό σύμφωνο το οποίο είναι ένα πρώτο συστατικό στοιχείο για αυτό το οποίο έλειπε για μια οικονομική ένωση η οποία θα έπρεπε να υπάρχει ε, για να λειτουργήσει σωστά η Ευρωζώνη. Και αυτό μετά μας οδήγησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την έκθεση Φανρόμπα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση που είναι απλά μια αρχή της ε, συζήτησης αυτής και πρέπει τους επόμενους μήνες να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συζήτηση. Και ξέρετε για να είμαι ειλικρινής δεν είναι σαφές αυτό για κανέναν το τι θα κάνουμε δηλαδή και δεν υπάρχει καν σαφήνεια για το ποια στοιχεία ε, μπορούν να γίνουν χωρίς αλλαγή της συνθήκης και ποια απαιτούν αλλαγή της συνθήκης. Παραδείγματος χάρη ξέρετε πως περισσότεροι έλεγαν στη συζήτηση πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην Τραπεζική Ένωση η οποία είναι εφικτή εντός των υφισταμένων συνθήκων και τα άλλα στοιχεία. Ίσως θα χρειάζεται να περιμένουν μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε, για να έχουμε μία νέα έκθεση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες δεν θα πάνε κατευθείαν προς Απλά θέλαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Οπότε σημειώνω αυτά τα οποία είπατε. Και βεβαίως πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των όσων γίνονται στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όσο γίνεται στο επίπεδο του Συμβουλίου. Και πράγματι είναι θεμητό αυτό, αυτή η ενισχύα του Κοινοβουλίου, γιατί για εμάς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βεβαίως ε, είναι ο προϊστάμενός μας, αλλά ε, δεν είναι ο δικός σας προϊστάμενος. Οπότε πρέπει να βρεθεί η θεσμική σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων και έχετε δίκιο και θα επανέλθω σε αυτό πως πράγματι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι νομοθέτης, ε, το γνωρίζουμε τώρα όλοι, ε, αλλά είναι ένα θεσμικό όργανο. Αλλά πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και ευχαριστώ βεβαίω ε, να επανέλθουμε όταν θα έχουμε περισσότερες πληροφορίε και όταν θα ξέρουμε πιο ξεκάθαρα πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα έχουμε μια συνέλευση, τι είδου τέτοια συνέλευση και τι εμπλοκή του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα έχουμε. Αλλά γνωρίζουμε όλοι πως η φιλοδοξία για εμάς, όπως είπα, είναι να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και οι πολίτες πιο κοντά στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει να βρεθούν τρόποι να κλείσει αυτό το κενό και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Πολλοί θα πούν πως δεν είναι τώρα η ώρα να γίνει μια συνέλευση, να επανεξετάσουμε τη συνθήκη, γιατί δεν θα περάσει μια καινούργια συνθήκη γιατί σε πολλές χώρες ε, υπάρχει τα λοιπά Αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Και γνωρίζουμε επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, να σκεφτούμε δηλαδή και εγώ ευχαρίστως να διαβάσω τις ε, εκθέσεις που προετοιμάζει η Επιτροπή σας για την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και την έκθεση Λαμασούρ επίσης. Γιατί γεγονός είναι και συνειδητοποιούμε όλοι πως ε, καταλήξαμε με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, σε έναν πολλαπλασιασμό των κέντρων εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μετά ακόμα και εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαμε μια σύνοδο κορυφής του Eurogroup που έλαβε χώρα ε, παράλληλα διαφορετικό θεσμικό όργανο αλλά τα αποτελέσματα του Eurogroup ε, ήταν υπό την αίρεση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά έχουμε την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο, νέο θεσμικό όργανο, την υπηρεσία της αυξημένες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν η οποία βεβαίω ε, θέλει να διαφυλάσει τις αρμοδιότητές της, την εκπεριτροπής Προεδρία. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ε, ρυθμιστεί καλύτερα αυτό το σύστημα το οποίο αυξάνεται και πληθύνεται. Νομίζω πως αυτός είναι μέρη ο ρόλος της εκπεριτροπής Προεδρίας να διασφαλίσουμε δηλαδή μια συνοχή και συνέργεια μεταξύ αυτών των κέντρων εξουσίας. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις σκέψεις μας από αυτόν και οτιδήποτε βεβαίω συνεισφέρει η Επιτροπή σας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά την προσχώρηση της Ένωσης στην ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Κύριε Ντάφ, Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περίμενε τη δική μου πίεση. Από ό,τι φαίνεται θα έρθουν και οι τελευταίες τους επιφυλάξεις. Αυτές είναι οι τελευταίες μας πληροφορίες. Οπότε οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξανανοίξουν και ελπίζουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο ζήτημα αυτό. Και βεβαίως σημείωσα τις παρατηρήσεις σας Κύριε Γκερέρα, σας ευχαριστώ για την στήριξή σας και για αυτό το οποίο είπατε για την πρώτη σας προεδρία, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ παρηγορητικό για εμάς, γιατί ξέρετε στα πιο δύσκολα ζητήματα δεν ξέρει κανείς που να θέσει τον πύχη. Αν το θέσει πολύ ψηλά δεν είναι σοβαρός, αν το θέσει πολύ χαμηλά χάνει την ευκαιρία να επιτύχει κάποια αποτελέσματα. Οπότε ε, εδώ πέρα βασιζόμαστε σε όλους σας να μας βοηθήσετε να πετύχουμε τη σωστή ε, ισορροπία. Και όπως είπατε στην περίπτωση μας ακόμη περισσότερο γιατί είμαστε μικρή χώρα, έχουμε κινητοποιήσει ολόκληρο το δημόσιο τομέα, όλους τους ανθρώπινους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και το κόστος αναλογικά είναι πολύ ψηλό για τη χώρα, αλλά αξίζει νομίζω να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και ξέρετε πως στις Βρυξέλλες είχαμε γύρω στα 90 άτομα, τώρα έχουμε πάνω από 200 για την Προεδρία. Επενδύουμε δηλαδή πραγματικά και κινητοποιούμε όλους τους πόρους μας. Και σημείωσα επίσης αυτό το οποίο είπατε για τον προπολογισμό του 2013 το Συμβούλιο χτες υιοθέτησε με ειδική πλειοψηφία την θέση του επί του προπολογισμού και θα έρθουμε τον Σεπτέμβριο να συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να ληφθεί πλήρως υπόψη αυτά τα οποία έπρεπε να ληφθούν πλήρως υπόψη. Τέλος, ε, τώρα για το δύσκολο ζήτημα της ε, διακυβέρνησης της Σέγγεν και ο κύριος Νταφ και ο κύριος Μέσερ Σμιτ ε, έθεσαν το σημαντικό αυτό ζήτημα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τα καλά νέα. καλά νέα είναι πως είμαστε σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χτες καταφέραμε να πείσουμε την Κορεπέρ να δεχτεί μια διαδικαστική πρόταση για να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ελπίζουμε αυτό να καταστεί δυνατόν τους ερχόμενους μήνες και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πέρα από το να σας διαβεβαιώσω πως θα εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά για να βρεθεί ένας τρόπος να προχωρήσουμε που θα σέβεται βεβαίως τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα βεβαίως υπάρχει άλλη πλευρά του θέματος που είναι πως ναι θεωρώ πως ο κύριος Μέσσερ Σμιτ έχει δίκιο, δεν πρέπει να κατηγορούμε την Προεδρία της Ίσως από πλευράς του εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχε, υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες ή θεωρούσε πως ε, η Προεδρία της Δανίας ε, δεσμεύτηκε για κάτι το οποίο δεν μπορούσε να κάνει αλλά και έτσι να είχαν τα πράγματα νομίζω πως ε, έδρασαν καλή την πίστη. Το πρόβλημα είναι βεβαίως πως δεν μπορούν να αλλάξουμε την νομική βάση παρά μόνο ομόφωνα σύμφωνα με δύο γνωμοδοτήσει τη νομική υπηρεσία του Συμβουλίου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν αυτό το οποίο λέει το Κοινοβούλιο, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι. Και νομίζω πω ο κύριο Ντάφ ήταν εκεί και γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ήταν εκεί όταν ε, συντάχθη το άρθρο 70, πως επέμειναν τα κράτη-μέλη στο ότι η Σέγγεν και τα σχετικά αυτά ζητήματα βασίζονται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και επέμειναν στην ιδέα αυτή του ελέγχου από τους ομολόγους. Οπότε όταν μιλάμε για την αξιολόγηση, μόνο για την αξιολόγηση. Τα κράτη-μέλη επέμειναν πως αυτό πρέπει να είναι αρμοδιότητα δική τους δεν θεωρούν πως αυτή η αρμοδιότητα είναι μια αρμοδιότητα η οποία έχει περάσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, αυτή είναι η άποψη των κρατών μελών και τελικά αυτό είπε και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου του τηλεχθέντος. Αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα όμως δεν είναι μια αξιολόγηση μόνο η αξιολόγηση είναι βεβαίως ε, ένα βήμα για κάτι άλλο και το πραγματικό ζήτημα εδώ πέρα είναι η διακυβέρνηση και το πώς θα επιτρέπουμε σε εξαιρετικές ε, περιστάσεις παραδείγματος χάρη την ε, επανεισαγωγή εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα κτλ. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε πως αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε τελική ανάλυση και εκεί. Εάν φύγει αυτό το καθαρά νομικό ε, στοιχείο του εάν ε, υπάρχει κάποια μεταφορά αρμοδιοτήτων ή όχι όσον αφορά την αξιολόγηση. Νομίζω πως για τα υπόλοιπα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ε, ξέρω πως ίσως κάποια κράτη-μέλη θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη νομική βάση για να αποφύγουν το να εμπλακούν. Αλλά σε τελική ανάλυση, <clears throat> αν μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ότι απλώς διαφωνούμε μοναχά σε αυτό το μεμονωμένο στοιχείο, ίσως για τα υπόλοιπα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με έναν τρόπο που είναι ικανοποιητικός και ξέρετε ότι η, η απόφαση του Συμβουλίου Εσωτερικών και Δικαστικών της 8ης Ιουνίου ήταν να μεταφερθεί μια σειρά αποζητήματα από την αξιολόγηση του κανονισμού στο μηχανισμό του κώδικα συμπεριφορά. Ναι, λοιπόν, επομένω πρέπει να δούμε ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα παραμείνουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών και ποια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απεπλεγμένο θέμα. Γνωρίζω ότι οι απόψει μα δεν είναι ταυτόσιμε κατά 100%, αλλά αν μπορέσουμε να επιτύχουμε επικάλυψη 95% νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα είναι κρίμα να μην προχωρήσουμε, διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλους μας και σε τελική ανάλυση και τώρα βγαίνω και από την εντολή μου ως Προεδρία πρέπει να σας πω ότι προσωπικά και η Κύπρος ως χώρα δεν χαίρονται για την ιδέα, δεν ενστερνίζονται την ιδέα του ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν μόνα τους και όποτε τους αρέσει να παίρνουν αποφάσεις για τα θέματα αυτά. Αλλά αυτό φυσικά ξεφεύγει από τη δική μου εντολή. Σας δίνω την προσωπική μου όμως οπτική γωνία για το θέμα αυτό στη συνέχεια. Για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Νταφ. Μακρηγορώ λιγάκι κύριε Πρόεδρε, σε πέντε λεφτά τελειώσω. Όπως έλεγα και στην αρχή, προσπαθώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής και απόλυτα έντιμος μαζί σας. Το άλλο θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Νταφ προκύπτει από αυτό το οποίο έγινε με τη διαδικασία για το δικαστήριο των ευρεσιτεχνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα θέμα του κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να έρθει και να ανατρέψει μία σχεδόν ηλυμένη απόφαση που είχε συμφωνηθεί μεταξύ, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μας όμως, είτε ακόμα και αν αυτό δεν έχει τυπικό χαρακτήρα, γιατί επισήμως είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο δίδει κατευθύνσεις προς το Συμβούλιο, ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο. Το Συμβούλιο αποτελείται, απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Όταν λοιπόν σας πούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάντε αυτό και εκείνο, αυτό είναι μια εντολή, δεν είναι μια απλή σύσταση. Κατανοώ λοιπόν ότι αυτό δημιούργησε ένα πραγματικό πρόβλημα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όταν πρόκειται για τη συμφωνία για τις ευρεσιτεχνίες, ξέρω ότι αυτό υπόκειται στη διαδικασία συναπόφασης και πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση μεταξύ των δύο σκελών της νομοθετικής εξουσίας. Αλλά και πάλι επειδή πρόκειται για ένα εγχείρημα στο οποίο έχουμε αποδηθεί και το οποίο έχει χρονίσει τόσο πολλά χρόνια, θέλω να σας κάνω μια έκκληση να είστε και εσείς στο, δυνατό, στο βαθμό του δυνατού πραγματιστές. Θα ήταν κρίμα να μην υπάρξει το ταχύτερο δυνατό μια συμφωνία τη στιγμή που οι επιχειρηματίες, οι βιομηχανικοί κύκλοι περιμένουν τόσο καιρό για να υπάρξει μια λύση στο θέμα αυτό και τώρα είναι σχεδόν έτοιμη αυτή η συμφωνία. Μπορεί να μην είναι ικανοποιητική αυτή η λύση κατά 100% αλλά ξέρετε όπως λένε οι Γάλλοι στο τέλος της ημέρας ότι το καλό είναι ο εχθρός του καλύτερου. Το καλύτερο μάλλον ο εχθρός του καλού. Καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η θέση σας, καταλαβαίνω την αντίδρασή σας και υπάρχει και ένα θέμα στο οποίο νομίζω κύριε Ντάφ εγώ νιώθω άνετα. Είναι ο αριθμός, ο καθορισμός του αριθμού των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να με ρωτήσετε εσείς, αλλά σας ξαναρωτάω εγώ, ποια είναι η κατάσταση των πραγμάτων. Η διαδικασία αυτή καθορισμού των αριθμών, του αριθμού των βουλευτών θα πρέπει να ξεκινήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά θα πρέπει να στείλετε τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μόνο τότε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει σε εσά για να σας ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη σας. Επομένως από εσά ξεκινάει η διαδικασία. Ξέρουμε ότι έχουμε περάσει τον αριθμό των 750 βουλευτών. Ξέρουμε ότι πρέπει το θέμα αυτό να επιληθεί πριν από τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, γιατί για την Κροατία δεν ξέρω αν θα είναι 11 ή 12 οι βουλευτές. Δεν ξέρω ακριβώς λοιπόν ποιος πρέπει να είναι ο σωστός αριθμός. Θα πρέπει να αναμείνουμε και αναμένουμε με αδημονία να υπάρξει η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον επανακαθορισμό του αριθμού των βουλευτών και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ως Προεδρία δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσω αυτό το θέμα. Συγχρόνως όμως <clears throat> είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και φυσικά ε, βρισκόμαστε εδώ για να εργαστούμε μαζί σας, για να ανταλλάξουμε απόψε ότι αν αυτό είναι απαραίτητο και φυσικά θα συνεργαστούμε μαζί σας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση για το θέμα αυτό. Για το ερώτημα του κυρίου Μπρόνς, <clears throat> ο οποίος αναφέρθηκε για το θέμα της Τουρκίας και της τουρκικής προσχώρησης. Τα είπατε όλα νομίζω κύριε Μπρόνς. Είναι δύσκολο για μένα επειδή είμαι Κύπριος να εμφανιστώ ως ε, κάποιος ο οποίος παίρνει μια συγκεκριμένη θέση για τα θέματα αυτά. Εμείς ως Προεδρία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως το δυνατόν πιο ουδέτερα και αμερόληπτα την Τουρκία. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να σας υπενθυμίσω τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου ότι δεν εναπόκειται στην Τουρκία να λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς να τακτοποιεί τα εσωτερικά της θέματα και πώς να λειτουργεί η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα άλλα, ως ε, Ευρωπαίος και πάλι ίσως ξεφεύγω από τις αρμοδιότητες μου ως Προέδρου του Συμβουλίου, ως ε, Ευρωπαίος και ως άτομο νιώθω προσβεβλημένος. Περισσότερο όμως σαν Ευρωπαίος παρά ως Κύπριος. Ως Κύπροι είμαστε απόλυτα συνηθισμένοι στο τμήμα του κόσμου που ζούμε να μην είναι τίποτα εύκολο να έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές από την Τουρκία. Ως Ευρωπαίος όμως θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανεχθούμε μια τέτοια συμπεριφορά, <clears throat> ιδίως όταν προέρχεται από μια χώρα που διεκδικεί την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία θα πρέπει να συμμερίζεται τις αξίες και τις αρχές μας και σε τελική ανάλυση θα πρέπει να κάνουμε κάτι για τη στάση της Τουρκίας. Σε σχέση με το ερώτημά σας, αν θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ή όχι, νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει αποφασιστεί στο παρελθόν όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Δεν εναπόκειται σε μένα να επικρίνω αυτή την απόφαση, αλλά εγώ κατανοώ ότι η λογική που προητάνευσε είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας για να ξεπεραστούν και κάποια προβλήματα, για να μπορέσει να βρεθεί και μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα, να περατωθεί η κατοχή ενός τμήματος της κυπριακής επικράτειας Βέβαια, εκ των υστέρων φαίνεται ότι η Τουρκία δεν, έχει, δεν είχε εκπληρώσει πλήρως τα προαπαιτούμενα της Κοπενχάγης, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ κοντά στο να επιτύχει την εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων. Τώρα είναι πέραν της εντολής μου αυτό, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από τότε, από την εποχή που υπήρξε η έναξη των διαπραγματεύσεων. για τον κύριο Μέσσερ Σμιτ για την έξοδο από την Ευρωζώνη και πιθανώς την έξοδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι όλοι μας προσπαθούμε να διαψεύσουμε το θέμα αυτό, την ύπαρξή του, μη γι' αυτό. Να το εξορκίσουμε. Θα ήταν πραγματικά άτυχο να προεδρεύει η Κύπρος την στιγμή κατά την οποία θα αντιμετωπιστεί μια τέτοια πιθανότητα. Πραγματικά δεν θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό και ελπίζουμε να μην συμβεί. Τώρα το αν υπάρχει κάποιο σενάριο τέτοιου είδους δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ίσως κάποιοι σκέπτονται το πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Και για το εάν η έξοδος από την Ευρωζώνη σημαίνει άμεσα έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το γνωρίζω. Νομίζω όμως ότι τελικά θα καταφέρουμε με έναν πραγματιστικό τρόπο να αποφύγουμε τέτοιου είδους σενάριοι αλλά δεν μπορώ να σας κατηγορήσω ότι κάνετε λάθος θέτοντας το θέμα. Και για την τελευταία παρέμβαση του κυρίου Κατσίνη, είμαι ευγνώμων πρόεδρε για αυτά που είπατε. Στα δικά μας τα μέρη στην Κύπρο έχουμε πραγματικά συνηθίσει να ζούμε και να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε εμείς να συνδυάσουμε τα διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό το κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επιτύχαμε να επιβιώσουμε κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και πλέον πρόσφατη περίοδος της ιστορίας μας δεν ήταν και από τις πιο λαμπρές όπως γνωρίζετε. Από την άλλη όμως θεωρούμε ότι οι εμπειρίες μας και οι γνώσεις μας για την περιοχή αυτή του κόσμου όπου ο ορθολογισμός δεν είναι η κυρίαρχη θα έλεγα αντίληψη μέσω όμως των εμπειριών μας θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και για την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις χώρες της Αραβικής Άνοιξης. Εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής εκτός από την Τουρκία όπως γνωρίζετε. Γνωρίζουμε τις χώρες αυτές και πιστεύουμε ότι αν μπορέσουμε να σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο και να τον αντικαταστήσουμε από ένα κύκλο εμπιστοσύνης, θα συνδυάσουμε τα κοινά στοιχεία και έτσι θα μπορέσουμε επιτέλους να αλλάξουμε την πλευρά αυτή του κόσμου, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίλυση και του Παλαιστινιακού και να βοηθήσει την μετάβαση προς τη δημοκρατία στη Συρία και να διασφαλίσουμε επίσης ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες και μεταρρυθμίσεις στις υπόλοιπες χώρες θα εξελιχθούν ομαλά προς μια δημοκρατική κοινωνία. Μέχρι τώρα για τις περισσότερες αραβικές χώρες της περιοχής δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως τι έχει συμβεί. Συνεργαζόμασταν με συγκεκριμένα καθεστώτα, τώρα έχουμε εκπλαγεί από τις εξελίξεις λίγο και πρέπει να βρούμε τον τρόπο χωρίς να παρέμβουμε στα εσωτερικά των χωρών αυτών να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Αν δεν το κάνουμε αυτό τότε έχω την αίσθηση ότι οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις θα γίνουν αντικείμενο κατάχρησης από ορισμένου που θα οδηγήσει σε απολυταρχικά καθεστώτα και ίσως και σε ισλαμικά καθεστώτα όχι λιγότερο απολυταρχικά από ό,τι μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει. Πρέπει να βοηθήσουμε για να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, ο σεβασμός των μειονοτήτων, η πολλαπλή επικοινωνία μας με την κοινωνία των πολιτών, με τους κοινωνικούς εταίρους, με τον επιχειρηματικό κόσμο και να εφαρμόσουμε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή την γνωστή ως more for more, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με το σωστό τρόπο με τις κυβερνήσεις της χώρες αυτές για να ανοίξει η κοινωνία τους και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των λαών της περιοχής που έχουν δίκαιες προσδοκίες και φιλοδοξίες για περισσότερη δημοκρατία. Αυτό που μπορώ να πω λοιπόν αυτό ήτανε Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μικρό άνοιγμα, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε την όθηση προς θετικές εξελίξεις. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν είναι εγγυημένο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα εν πολλής στις ε, ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής σας. Εγώ ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Μαυρογιάννη για τις απαντήσεις σας. Εμείς εκτιμήσαμε δεόντως αυτά τα οποία είπατε, εγώ εξετίμησα δεόντως αυτά τα οποία είπατε και τον έξυπνο τρόπο με τον οποίο μπορέσατε να συνδυάσετε τις προσωπικές σας πεπιθήσεις με την απαραίτητη βέβαια προσοχή επιφυλακτικότητα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει έναν διπλωμάτη. Καταλάβαμε όμως τον τρόπο που σκέπτεστε, καταλάβαμε τις επιθυμίες σας και ε, ευχόμαστε εγκαρδίως η Κυπριακή Προεδρία να σταθεί παράγωνα ανάπτυξης, ευημερίας, εμπιστοσύνης και ελπίδας. Όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και την δική σας χώρα και την δύσκολη κατάσταση στην περιοχή σας. Ό,τι καλύτερο λοιπόν. Μια Μιας και προετοιμαζόμαστε για τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να σας ενημερώσω λίγο για τη συνάντηση των συντονιστών που έγινε χθε το απόγευμα. Κατά πρώτον, και σας τα μεταφέρω αυτά φυσικά για να εγκρίνετε στο σύνολό σας ε, τις αποφάσεις αυτές για την πρόταση τροποποίησης του άρθρου 49 αποφασίστηκε η απόφαση αυτή, η πρόταση αυτή να ενταχθεί σε μια μελλοντική ευρύτερη έκθεση που να περιλαμβάνει και άλλα άρθρα του κανονισμού. Και αυτό γιατί η διάσκεψη των Προέδρων θα κάνει μια ακρόαση, ένα σεμινάριο γύρω από το θέμα αυτό και περιμένουμε και εκθέσεις για τα άρθρα 48, 50, 20 και 27 του κανονισμού για την ερμηνεία του 187 και του 191 στην επόμενη συνεδρίασή μας θα σας προτείνω ένα σχέδιο επιστολής για την έκθεση της ε, ε, Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών για την Ουγγαρία είναι απαραίτητο και η Επιτροπή μας να εκφέρει μια γνωμοδότηση. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ε, ο εισηγητής μας θα είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα εξετάσει ο εισηγητής αν θα εκδώσει μια γνωμοδότηση ε, στην πρώτη φάση ή στη δεύτερη φάση ή και στις δύο. Ξέρετε ότι Μέχρι το 2013 έχουμε ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα σε σχέση με τη διαδικασία αυτή και θα, δει, θα εκτιμήσει ο εισηγητής. Τώρα για την πορεία προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση, ο εισηγητής θα οριστεί από πλευρά της σοσιαλιστική ομάδα. Αυτή είναι η πρόταση των συντονιστών. Θα εξετάσουμε τους τρόπους συνεργασίας με την Επιτροπή ΕΚΟΝ και προτείνεται να γίνει και μία μικρή συνάντηση των συντονιστών των δύο αυτών επιτροπών την πρώτη εβδομάδα, τις πρώτες εβδομάδες του μηνός Σεπτεμβρίου. Θα προσκαλέσουμε επίσης και έναν εκπρόσωπο της Προεδρίας για να εκφραστεί σε σχέση με τις εκθέσεις που προανέφερα. Για την ΣΕΝΤΕ η γνωμοδότηση θα γίνει από Πλευρά των φιλελευθέρων, ο κύριος Νταφ. Για τη σύνθεση του δικαστηρίου, η συγητής για γνωμοδότηση θα είναι από την ομάδα της Ευρώπης των Εθνών και θα είναι μάλλον ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, νομίζω ότι θα είναι ο κύριος Τσαρκόφσκι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για το θέμα των πολιτικών ευρωπαϊκών κομμάτων. Ο εισηγητής θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει δύο σημεία, δύο πόντους η έκθεση αυτή, θεωρείται πολύ σημαντική, γιατί ασχολείται και με τα θέματα της χρηματοδότησης των πολιτικών ευρωπαϊκών κομμάτων και ανάλογα για το αν θα δοθεί επί της ουσίας ή επιγνωμοδοτήσει η συγκεκριμένη αυτή έκθεση στην Επιτροπή μας θα δούμε πόσο θα κοστίσει σε εισαγωγικά. Για την οργάνωση ακρόαση στη συμμετοχική δημοκρατία από πλευράς του κυρίου Χέφνερ είναι δεκτή η πρόταση αυτή, θα διεξαχθεί αυτή η ακρόαση. Σχετικά με το αίτημα του κυρίου Νταφ για να δημιουργηθεί μια ακρόαση ή μια ομάδα εργασίας ή ένα σεμινάριο για το θέμα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι μπορούμε να δεχθούμε την διοργάνωση αυτής της ακρόασης, ίσως να γίνει όμως το 2013 γιατί θα πρέπει νομίζω να περιμένουμε και την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια θα επιμείνει να αποκτήσει την γνωμοδότηση αυτή. Δεν έχουμε άλλες παρατηρήσεις, εφόσον δεν διαφωνείτε, αυτά που σας είπα γίνονται δεκτά. Και περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε τρεις εκθέσεις. Η πρώτη είναι η έκθεση Hefner για τη σύναψη μιας διοργανικής συμφωνίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την μετάδοση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές από πλευράς του Συμβουλίου και που άπτονται της πολιτικής ασφαλείας και της πολιτικής ε, ε, στον τομέα των διεθνών σχέσεων. Λοιπόν, υπάρχει μια τροπολογία, η τροπολογία 3 του κυρίου Γκουερέρο. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Ένας εκφράζεται κατά. Γίνεται δεκτή. Θέτω σε ψηφοφορία τώρα την τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη Β του κυρίου Γκουερέρο. Ποιοι είναι υπέρ της 1. Κατά. Ο κύριος Νταφ διαδικαστικό. Μια ερώτηση για τροπολογία 2 του κυρίου Γκερέρο που κάνει λόγο για συνθήκες και άλλα νομικά κείμενα. Κάπως μυστηριώδης διατύπωση. Δεν χρειάζεται τόσο μυστήριο. Εγώ θα προτιμούσα να φύγουν αυτές οι λέξεις από εκεί, εάν συμφωνεί και ο κύριος Γκερέρο. Για να είναι σαφές το σε τι αναφερόμαστε. Ευχαριστώ. Αναφέρεστε στην τροπολογία υπαρίθμου 2, κύριε Νταφ. Ας ακούσουμε την άποψη του κυρίου Γκουερέρο. Συμφωνείτε με αυτά τα οποία προτείνει ο κύριος Νταφ. Ψηφίζουμε λοιπόν με την παρατήρηση του κυρίου Νταφ. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή η τροπολογία. Θα ψηφίσουμε τώρα την τροπολογημένη πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή ομόφωνα. Συγχαρητήρια κύριε Χέφνερ ομόφωνα. Α, κάποιος ε, διαδικαστικό, κύριος Φόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις αρχικές σας παρατηρήσεις είπατε πως θα ψηφίσουμε τρία θέματα. Από όσο ξέρω το ζήτημα του πρωτοκόλλου της Τσεχίας ακόμα ε, προβλέπεται να ψηφιστεί. Το συζητήσαμε χτες, είπανε ΕΛΚ και οι σοσιαλδημοκράτες πως δεν θένε να το ψηφίσουμε, αλλά δεν έχει αποφασίσει κάτι τέτοιο η Επιτροπή. Εάν έχει ληφθεί απόφαση να μην ψηφιστεί, παρακαλώ να το ανακοινώσετε και να κάνει και ένα συνάδελφος πιθανώς μια πρόταση να μην ψηφιστεί. Yes, no, I'm, sorry that Mr. Fox does not remember exactly. Λυπούμε γιατί ο κύριος Φόξ δεν θυμάται τι έγινε χτες. Χτες αποφασίσαμε το ότι ο πρόεδρος σημείωσε πως υπήρχε μια ευρεία πλειοψηφία υπέρ της αναβολής. Ανακοίνωσε αυτή την απόφαση, κανείς δεν είχε αντίρρηση, η απόφαση ληφθεί. αυτό έγινε όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση και καθορίσαμε την ημερήσια διάταξη. Δεν μπορεί να ξαναλλάξει τώρα. Κύριε Πρόεδρε, ε, δεν συνέβησαν αυτά χτες. Έγινε μια γενική συζήτηση και ο κύριος Νταφ και εγώ είπαμε πως δεν συμφωνούμε με αυτό. Δεν έγινε ψηφοφορία. Το θέμα υπάρχει ακόμα στη μερίσια διαταξία. Αν ο κύριος Γκουαλτιέρη θέλει να, να διαγραφεί, ευχαριστώ. Ma Συγγνώμη, παίρνω το λόγο γιατί σαν πρόεδρος έχω καθήκον να σημειώσω με σωστό τρόπο αυτά τα οποία έγιναν. Ακούσαμε τις γνώμες όλων, είπαμε ότι οι δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες ζήτησαν την αναβολή της ψηφοφορίας σε σχέση με την Τσεχία και ο εισηγητής είχε δεκτεί είχε κάνει δεκτή αυτή την πρόταση. Δεν είχαμε κάνει επίσημη ψηφοφορία, είχαμε πει, είχα δηλώσει εγώ ότι θα αφαιρεθεί το θέμα από την ημερήσια διάταξη γιατί υπήρχε μια προφανής πλειοψηφία. Αυτά έγιναν χτες. Για τα θέματα της ημερήσια διάταξης εγώ είμαι υπεύθυνο και έτσι έγιναν τα πράγματα. Ο κύριος Ντάφ έχει ζητήσει το λόγο. Κοιτάξτε, πριν από οτιδήποτε άλλο προσπαθώ να είμαι ρεαλιστής και είναι ξεκάθαρο ότι οι σοσιαλιστές και οι χριστιανοδημοκράτες ήσαν χθε κατά της σημερινής ψηφοφορίας. Είπα παρόλα αυτά χθε ότι αν υπάρξει αναβολή, η αναβολή θα οριστεί μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο. Όχι γενικά γιατί πρέπει το Κοινοβούλιο να πάρει μία απόφαση πάνω σε ένα σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Αν θέλετε εσείς να ρυθμίσετε με πιο τακτικό τρόπο την απόφαση αυτή, μπορούμε να πάρουμε μία επίσημη ψήφο, αν θέλετε, να γίνει μία ψηφοφορία. I can only say όπως χθες συμφωνήσαμε με το δικό σας το αίτημα περί αναβολής. Μπορώ να το πω και σήμερα, αλλά το συμφωνήσαμε και χθες. Για μένα έχει λήξει το ζήτημα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές ότι τα πράγματα έγιναν όπως είπε ο κύριος Νταφ. Δεν αποφασίζουμε να μην αποφασίσουμε, αλλά να παραπέμψουμε το θέμα για τον μήνα Σεπτέμβριο. Συμφωνείτε παρακαλώ. Αν θέλετε εσείς να ξαναψηφίσουμε, γιατί όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό συνέβη χθε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα που είναι το εξής. Χθε ήταν σαφές για όλους ότι υπήρχε αυτή η αναβολή. Και εμείς ως συνάδελφοι στην Επιτροπή αυτή θα πρέπει να συζητάμε μεταξύ μας καλή την πίστη ο κύριος Φόξ και ο κύριος Μπρόντς ξέρανε πολύ καλά ότι είχε υπάρξει αυτή η αναβολή. Είναι ένας τεχνητός ελιγμός μονάχα για να πούνε κάτι διαφορετικό. Εγώ πράγματι απογοητεύομαι. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η συμπεριφορά τους σαν Βρετανών κοινοβουλευτικών θα έπρεπε να ήταν ένα υπόδειγμα για όλους τους δημοκράτες. Εάν λοιπόν λειτουργείτε καλή τη πίστη, δεν πρέπει να κάνετε αυτούς τους μικροπολιτικούς ελιγμούς εδώ. Είναι σαφές, ήταν απόλυτα σαφές ότι είχαμε αποφασίσει να αναβάλουμε την ψηφοφορία και δεν ψηφίζουμε για όλα τα πράγματα. Πολλές φορές υπάρχει απλώς η συμφωνία των συντονιστών. Και νομίζω ότι ο Φόξ κατανοεί ότι όταν κάνουμε την κατανομή των εκθέσεων δεν ψηφίζουμε. Όταν υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ μας είναι συμφωνία. Και απλώς καταγράφεται η συμφωνία μας από τον πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα τώρα να ψηφίσουμε, πέραν του ότι θα υποσκάψουμε τις αποφάσεις των συντονιστών και θα αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια του πρόεδρου μας. Πιστεύω λοιπόν ήταν σαφής η χθεσινή απόφαση και δεν έχει κανένα λόγο να την αμφισβητήσουμε τώρα. <clears throat> Ο κύριος Μπρόντς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές, ήταν σαφές ότι το ΕΛΚ ήθελε να γίνει η αναβολή. Ήταν σαφές ότι και οι σοσιαλιστές ήθελαν να αναβληθεί αυτή η ψηφοφορία και συμφώνησε και ο εισηγητής. Δεν υπήρξε καμία πρόταση αναβολής, ούτε καν απόφαση. Τότε δεν χρειάζεται να πάμε στην Ολομέλεια, απλώς να ζητήσουμε από το ΕΛ και τους σοσιαλδημοκράτες να μας πούν τι θέλουν και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάτι στην Ολομέλεια, μπορούμε να καθόμαστε στα γραφεία μας και να περνάμε με ζάχαρη. Ο κύριος Κόξ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για να διορθώσω τον κύριο Τρασκόφσκι. Το θέμα αυτό δεν εξετάστηκε από τους συντονιστές. Εξετάστηκε από την Επιτροπή μας ως σύνορο. Είναι απόλυτα σαφές σε μένα το αν θα προχωρούσε η ψηφοφορία για το τσεχικό πρωτόκολλο ή όχι, αυτό υπήρξε συζήτηση στην Επιτροπή μας και με υποστηρίζει ο Άντριου Νταφ, όχι στους συντονιστές. Εγώ κατανοώ ότι είμαι σε μειοψηφία, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Όταν είμαστε σε μία επιτροπή, δεν αρκεί να πούν οι δύο μεγάλες ομάδες ότι θέλω να υπάρξει μία αναβολή και ότι αυτό σημαίνει δεν χρειάζεται να υπάρξει συζήτηση και ψηφοφορία. Δεν παίζω μικροπολιτικά παιχνίδια. Απλώς θέλω να καταγραφεί σήμερα ότι η ομάδα μας ήθελε να γίνει αυτή η ψηφοφορία σήμερα. Τώρα έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Ξέρω ότι τα εκατομμύρια των πολιτών που μας παρακολουθούν από το ίντερνετ θα το σημειώσουν και αυτοί με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ψηφοφορία σήμερα, αλλά έχουμε καταγράψει τη θέση μας. Αλλά καταγράφω και τη δική σας δήλωση, το θέμα αυτό θα επανέλθει το Σεπτέμβριο και χαίρομαι που και αυτό καταγράφεται πια στα πρακτικά ο κύριο Χέφνερ και μετά θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ωραία είναι το γεγονό ότι καταγράφονται οι συνεδριάσεις μα. Είναι θέμα δημοκρατία και διαφάνεια. Αλλά κάπω περιπλέκονται τα πράγματα και γίνονται παράξενα αν εμεί δεν μιλάμε μεταξύ μα, αλλά μιλάμε προ το κοινό και το υπερπέρα. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά πρέπει να επιλύονται στην Επιτροπή μα. Γι' αυτό μα εξελέξαν. Το θέμα αυτό συζητήθηκε χθε. Ζήτησε το ΕΛΚ αναβολή, ζήτησε η σοσιαλιστική ομάδα αναβολή. Εσείς είπατε να μην γίνει αναβολή, εμείς είπαμε να γίνει αναβολή και επομένως καταλήξαμε στο ότι θα γίνει αυτή η αναβολή γιατί υπήρχε μια σαφής ε, πλειοψηφία υπέρ της αναβολής. Τώρα το να παίζουμε παιχνίδι αυτό δεν μου αρέσει. Κοιτάξτε, ας κλείσουμε το θέμα τώρα, ας μην χάνουμε άλλο χρόνο. Θα βάλουμε στα πρακτικά αυτά τα οποία έτσι και αλλιώς ακούστηκαν και τις δηλώσεις του κυρίου Φόξ. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία επί της εκθέσεως Τσαρκόσκη για την τροποποίηση του άρθρου 123 του κανονισμού σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις και του άρθρου 42 σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, πρώτη συμβιβαστική τροπολογία Αλφα κεφαλαίο, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Α, κάποιος θέλει το λόγο, κύριος Νταφ. Πρόεδρε, εγώ έχω, αντί... εγώ έχω αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Bene, allora, data l'opposizione... Κοιτάξτε, μια και υπάρχει αντίρρηση από ένα μέλο, δεν θα ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε όμω τη συμβιβαστική ω είχε. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. αποχέ. Δεκτή. Η συμβιβαστική. Κλείνει το μικρόφωνο του πρόεδρος. Λοιπόν, υπάρχει εδώ κατά διέρεση ψήφος που έχει συζητηθεί από τους πρασίνους. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. αποχές δεκτό. Συμβιβαστική τροπολογία καλύπτει λοιπόν τις υπόλοιπες τροπολογίες μέχρι την 53. Περνάμε τώρα στη δεύτερη συμβιβαστική, ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Δεκτή και η δεύτερη συμβιβαστική, ομόφωνα και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε απευθείας στην τροπολογία 3 του εισηγητή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Έπεται η 58. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 59 του κυρίου Νταφ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 60 το δεύτερο τμήμα μάλλον της τροπολογίας 60, 60 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 61 έχει καταπέσει. Περνάμε στην 62 Σόλτς. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 έχει αποσυρθεί, 64 έχει αποσυρθεί, περνάμε στην 65. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η 4 του εισηγητή ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεν θα ψηφίσουμε την 67 γιατί έχει καταπέσει 4, έχει γίνει δεκτή η 4. Ο κύριος Νταφ, διαδικαστικό, μάλλον να διευκρινίσω κάτι. δεν μπορέσαμε εμείς σαν Επιτροπή να τροπολογήσουμε τις προτάσεις για το άρθρο 42, γιατί χάσαμε τις προθεσμίες, νομίζω ότι εμείς στη φιλελεύθερη τουλάχιστον ομάδα θα θέλαμε να γίνει δεκτή η τροπολογία μας στην Ολομέλεια επί του άρθρου 42 και γι' αυτό θα θέλαμε να ζητήσουμε και από τη διάσκεψη των Προέδρων να το συζητήσει το θέμα στην Ολομέλεια παρακαλώ. Η έκθεση δηλαδή αυτή για το 42 να συζητηθεί στην Ολομέλεια πριν την ψηφοφορία. Καλώς. Συμβιβαστική η 3, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 68 καλύπτεται από τη συμβιβαστική. Περνάμε στην 39 γκούρμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Η 42 τώρα. 42. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 40 έχει πλέον καταπέσει λόγω της υιοθέτησης της 42 και το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία 41. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ της 5. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Γκουρμαϊ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8. Ταυτόσημη με την 7. Οπότε δεν την ψηφίζουμε. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 12 είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά απορρίπτεται. Φτάσαμε στην συμβιβαστική D του εισηγητή, καλύπτει από τη 19 μέχρι την 21 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Πηγαίνουμε τώρα απευθεία στην τροπολογία 22. Α, για μια στιγμή. Κατάλαβα, λέει ο πρόεδρος, πηγαίνουμε τότε στην επόμενη συμβιβαστική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα πηγαίνουμε στην F. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία, όλες οι άλλες έχουν καταπέσει. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δύο είναι κατά. Αποχές. 17 υπέρ, 2 κατά λοιπόν. Καλώς. Και φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία, την έκθεση Μέσερ για την 28η ετήσια έκθεση για, την, για τον έλεγχο εφαρμογής του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την τροπολογία 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 Ραντζέλ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 4 Ραντζέλ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 5 γκουρμάι και τα λοιπά υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 6 έφνερ υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 αρανχέλ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 14 Ρέγνερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οι 11 και οι 13 καταπίπτουν. 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται η 15. Ψηφίζουμε την 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Καταπίπτει λοιπόν η 17 και η 18. Παραμένει η 19. Ποιοι είναι υπέρ της 19. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τελική ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Λοιπόν, ευχαριστώ τους ε, εισηγητές. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο. Ευχαριστώ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 Έχουμε στην ημερήσια διάταξη πριν από το θέμα το σημαντικό τη διακυβέρνηση την πολυεπίπεδη έχουμε και το σημείο 16 το οποίο αφορά την ενδιάμεση έκθεση ε, για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε σχέση με την διαδικασία έγκρισης του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Ο κύριος Τσαρκόφσκι είναι ο εισηγητής.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 Allora, eh, Καλώς. Ο συνάδελφος Τσακόσκι μας είπε ότι θα προτιμούσε το άρθρο 16 της ημερήσιας διάταξης, την ενδιάμεση έκθεση και τα λοιπά της διαδικασίας έγκρισης δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου 2014-2020, ότι προτιμά την αναβολή και θα αναφερθούμε τώρα στο πιο συγκεκριμένο θέμα, στο πιο σημαντικό θέμα, το 17, συνταγματικά θέματα που τίθενται στα πλαίσια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, έκθεση Τσαρκόφσκι Τσαρκώσκι-Γουαλτιέρη αλλά είναι εδώ ο κύριος Γουαλτιέρη Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλος ιδιαιτέρως τον καθηγητή κύριο Μαντούρο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Εγώ σαν πρόεδρος ε, το εκτιμώ δεόντως, το γνωρίζω πολύ καλά, έχω ήδη συναντηθεί με τον καθηγητή Μαντούρο, είναι εμπειρογνώμων στο συνταγματικό δίκαιο, έχει μια, ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό και τον ευχαριστώ που ήρθε εδώ. Ευχαριστώ και όσους οργάνωσαν πολύ ε, σύντομα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την συνάντηση αυτή. Θα ακούσουμε πρώτα την γνωμοδότηση του κυρίου Μαντούρο και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λείψω, αλλά θα με αντικαταστήσει ο κύριος Μέσερ Το Ο κύριος Γκουαλτιέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Μαντούρο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να επαναλάβω τις βασικές γραμμές της εκθέσεως ε, στην οποία έχω ήδη αναφερθεί. Εδώ ήρθαμε να ακούσουμε κυρίως τον κύριο Μαντούρο και να συζητήσουμε μαζί του. Νομίζω όμως, και το λέω αυτό πολύ συνθετικά, ότι μπορούμε να παρουσιάσουμε με συγκεκριμένο τρόπο το θέμα το οποίο εμείς είχαμε ορίσει σαν αντικείμενο της έκθεσής μας και το οποίο αν δεν κάνω λάθος επιβεβαιώθηκε και από τις περαιτέρω θα έλεγα υποθέσεις τις οποίες έπρεπε να μας, οι οποίες έπρεπε να μας απασχολήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε εμείς μια έκθεση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ένα θέμα το οποίο είχαμε προτείνει να ορίσουμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο, επί τη βάση τριών βασικά ασυμμετριών, τριών στοιχείων. Εν πάση περιπτώσει το χαρακτηριστικό το πολυεπίπεδο δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το θέμα είναι οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωζώνη, η ασυμμετρία ανάμεσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ασυμμετρία που υπάρχει στον τομέα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τα κράτη-μέλη και η ασυμμετρία ανάμεσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υποχρεώσεις τους και τις ρυθμίσεις τις διακυβερνητικές όπως το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τα υπόλοιπα δύο ταμεία. Λοιπόν, αυτές τις δύο μορφές, τις τρεις μορφές ασυμμετρίας είναι κάτι το οποίο οφείλεται ε, και σε κάποιες οικονομικές πραγματικότητες αλλά και ε, στο λεγόμενο δημοκρατικό έλλειμμα. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα ουσίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι η συμμετρία ανάμεσα στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα νομισματικά και στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών τις οποίες ορίζει αντικείμενο της διακυβερνητικής διάστασης η ίδια η συνθήκη και αυτό είναι κάτι το οποίο περιπλέκει θα έλεγα το πλαίσιο μέσα στο οποίο κατανέμονται ε, οι πόροι όπως ξέρετε το 99% του ΑΕΠ στα κράτη-μέλη και το 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι ότι εδώ τίθεται βέβαια και το θέμα των ελλημάτων, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν θα απασχολήσει τον κύριο Μαντούρο. Υπάρχει και η παρουσία συμμετρικών σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς. Εδώ τίθενται και θέματα νομιμοποίησης όπως και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οφείλουμε να εξετάσουμε και υπάρχει τέλος και ένα βαθύτατα πολιτικό θέμα στα πλαίσια του δημοκρατικού ελλείμματος όπως λέμε που παράγει συνεχώς εντάσεις διότι η κρίση ενίσχυσε κατά κάποιο τρόπο την σχέση της διακυβέρνησης στο εσωτερικό της δημοσιονομικής πειθαρχίας μέσω των ρυθμίσεων του ΠΑΚ και pack. Αν δεν υπάρξει μια παράλληλη αναπροσαρμογή, μια ενίσχυση δηλαδή της διακυβέρνησης, της εσωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι της εφαρμογής της πολιτικής αυτής σε εθνικό επίπεδο, Όλα αυτά είναι θέματα, εν πάση περιπτώσει, που θα πρέπει να εξετάσουμε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης σε τρία επίπεδα. Πρώτον, να θέσουμε τα προβλήματα. Δεύτερον, να δούμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η συνθήκη. Αυτό που λέει ο καθηγητής Μαντούρο, συνταγματικές αλλαγές χωρίς τροπολογίες της συνθήκης και δεύτερον πιθανές αλλαγές στη συνθήκη που θα πρέπει να, θα έλεγα, να έχουμε υπόψη μας σε μια τρίτη φάση. Και υπάρχουν και αρκετά άλλα επιμέρους θέματα τα οποία θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Το άρθρο 126, ο συνδυασμός του 126 με το 152, η ενισχυμένη συνεργασία, το εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομιμοποιείται πλήρως και στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωζώνης. Ξέρετε ότι ο πρώτος κανονισμός θα ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο από 27 χώρες, γιατί από 27 αποτελείται το Κοινοβούλιο, ενώ το Συμβούλιο στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελείται από 17 χώρες στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Και υπάρχει και το θέμα της διαδικασίας του Σέγγεν που είναι περισσότερο πολιτική διαδικασία παρά θεσμική. Και όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια περαιτέρω πολιτικοποίηση των ευρωπαϊκών οργάνων και εδώ τίθεται το θέμα των πολιτικών κομμάτων και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τέλος, περιπλοκότατο θέμα, το θέμα του προϋπολογισμού, οι διαδικασίες εδώ είναι πολύ περίπλοκες, ο καθορισμός των ιδίων πόρων, ο καθορισμός του ελαχίστου επίπεδου για το MFF, όπως επίσης και η ιδιαίτερη θέση την οποία κατέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της προσπάθειας επιβολής αντιπροσώπευσης χωρίς φορολογικές ρυθμίσεις ή των φορολογικών ρυθμίσεων χωρίς πολιτική αντιπροσώπηση. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά σας τα λέω λιγάκι σχηματικά, αλλά παρόλα αυτά αυτά είναι τα πλαίσια των θεμάτων τα οποία ορίσαμε μέχρι τώρα σαν θέμα ουσίας θα έλεγα για να συζητήσουμε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Γουαλτιέρη. Το λόγο έχει ο κύριος Τσαρκόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε το γενικό πλαίσιο το οποίο έχει και δεν θέλω να καταπανίσω περισσότερο χρόνο. Νομίζω ότι η συζήτηση για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ε, είναι κάτι που μας απασχολεί εδώ και πολύ χρόνο. Από τη δεκαετία του 70, αλλά πιο έντονα από τη δεκαετία του 90 και μετά, και <clears throat> μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να πάρουμε πολλές σημαντικές αποφάσεις για το πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε σχέση με τις συνθήκες, παρά το γεγονό ότι δεν υπάρχει ακόμα μια σαφής οροθετική γραμμή και είναι δύσκολο να εξηγήσουμε ότι είναι πραγματιστική αυτή η αντιμετώπιση στους εκλογείς μας. Είναι δύσκολες βέβαια οι στιγμές που διερχόμαστε λόγω της κρίσης, αλλά και σε ό,τι αφορά τη θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η συνθήκη του Λισαβόνας υπετίθεται ότι θα δημιουργούσε μεγαλύτερη σαφήνεια για αυτά τα θέματα, αλλά σε κάποια από αυτά, ιδίω σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί η συνθήκη για να γίνει πιο αποτελεσματικός ο λόγος μας στα θέματα αυτά, ιδίω όταν πρόκειται για το ρόλο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα σε σταυροδρόμι. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαφυλάξουμε το ευρώ και κάποιοι βέβαια δεν συμφωνούν με αυτή την άποψη γιατί συγχρόνως Θέλουμε να σώσουμε και το ευρώ, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε και τη θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρώπης και την σαφήνεια της θεσμικής αυτής αρχιτεκτονικής και την ενωσιακή μέθοδο και να αποφύγουμε να υπάρξει μια μορφή ρηγματοποίησης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία μπορεί να είναι μόνιμη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό που έχουμε ένα εμπειρογνώμονα ο οποίος μπορεί να μας παρουσιάσει αυτά τα θέματα. Έχουμε την ευκαιρία αυτή να ακούσουμε και όχι απλώς να συζητάμε μονάχα. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι μπορούμε, τι δυνατότητες μας δίνει το τωρινό πλαίσιο των συνθήκων, χωρίς να προχωρήσουμε σε περαιτέρω ριζοσπαστικές αλλαγές και πώς να προχωρήσουμε χωρίς να υπονομεύσουμε τις δομές που έχουμε ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι να ξαναγυρίσουμε σε προτάσεις όπως αυτές που διατυπώθηκαν στη δεκαετία του 60 να αλλάξουμε τελείως τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην προχωρήσουμε λοιπόν σε κάποιες διακυβερνητικές συμφωνίες που θα αλλάξουν το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο λοιπόν γινόντουσαν διαπραγματεύσεις για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, η θέση μας ήταν αυτή. Από την πλευρά του Κοινοβουλίου να διατηρήσουμε το πλαίσιο του Κοινοβουλίου και αν πρέπει να δεχτούμε κάποιες διακυβερνητικές λύσεις να τις σχηματοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε εν καιρό να μπορούν να συμπεριληφθούν στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σώσουμε λοιπόν το ευρώ χωρίς να καταρακώσουμε τα επιτεύγματα των τελευταίων 50 ετών και να μην οδηγηθούμε σε κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνω το λόγο λοιπόν στον καθηγητή Μαδούρο. Σβήνουμε τα φώτα και τον ακούμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για την πρόσκληση να έρθω εδώ. Και να πω πως όπως αναφέρθηκε, πολλές από τις προτάσεις και την ανάλυση που θα κάνω τα επόμενα 15-20 λεπτά προσπαθούν να σκεφτούν πιθανέ συνταγματικές αλλαγές για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Αλλά χωρίς οπωσδήποτε να απαιτηθεί αλλαγή της συνθήκης. Επίσης, θα ήθελα να κάνω άλλη μία υποσημείωση, όπως ίσως αντιληφθείτε τα επόμενα 15-20 λεπτά, πολλές από τις προτάσεις που κάνω σχετίζονται με τη δομή των πολιτικών της Ένωσης. Και αυτό σχετίζεται με το ότι και οι συνταγματικές αλλαγές απαιτούν αλλαγή της συνθήκης, αλλά, οι θεσμικές αλλαγές, αλλά και γιατί προσπαθώ να τονίσω εδώ και πολλά χρόνια πως η δημοκρατική νομιμοποίηση της διακυβέρνησης Ένωσης σχετίζεται και με την δομή των πολιτικών της, με το πώς επικοινωνεί με τους πολίτες της, αλλά και βεβαίως από τις θεσμικές αλλαγές. Ελπίζω να γίνει σαφές αυτό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μοιράσω την παρέμβασή μου σε δύο μέρη. Το πρώτο θα προσπαθήσει να θέσει τις τωρινές προκλήσεις διακυβέρνησης στο πλαίσιο της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το κάνω γιατί θεωρώ πως είναι σημαντικό. Αρκετό κομμάτι της ανάλυσης κρίσης ε, αφορά την οικονομική διάσταση της και εγώ θα ήθελα να κάνω μία ανάλυση της δημοκρατικής πτυχής ναι, δεν μιλάμε μόνο για τις ε, δημοκρατικές ε, και τις απαντήσεις που δόθηκαν στην κρίση, αλλά και το ποιε είναι οι αποτυχίες της δημοκρατίας που οδήγησαν σε αυτή την κρίση, γιατί νομίζω πως μόνο εάν αντιληφθούμε τη δημοκρατική διάσταση στη βάση της κρίσης και τις δυσκολίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να απαντήσει αυτή την κρίση, μόνο έτσι, κατά την άποψή μου, θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε καλύτερα το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά τις ε, νέες ε, δομές διακυβέρνησης και τον τρόπο νομοποίησής τους. Οπότε το ευρώ σε ένα μεγάλο βαθμό είναι μία απάντηση στην αυξανόμενη αλληλεξάρτηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επίσης αυξάνει και την αλληλεπίδραση εντός του. Και αυτό το οποίο νομίζω καθιστά σαφές αυτή η κρίση είναι πως δεν έχουμε αντιληφθεί αυτή την αλληλεξάρτηση. Και αυτό είναι μια αποτυχία της δημοκρατίας. Δεν έχουμε αντιληφθεί τον βαθμό των δημοκρατικών αλλαγών που έχουν γεννήθει και δημιουργηθεί από αυτή ήταν την αλληλεπίδραση. Και θα έλεγα πως έχουμε δύο είδη δημοκρατικής λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τις οποίες δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει. Το πρώτο, ένα αφορά τις ε, αυξημένε ε, δημοκρατικές εξωτερικότητες. Παραδείγματος χάρη με την αυξημένη ολοκλήρωση υπήρχαν πιθανές αρνητικές εξωτερικότητες σε άλλα κράτη. Και αυτό είναι πρόβλημα, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη τη προβλήματα άλλου κράτους στην εσωτερική δημοκρατική διαδικασία. Αλλά και εδώ πέρα υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα της δημοκρατικής λειτουργίας, δηλαδή την αδυναμία ρύθμισης ε, των ε, υπερεθνικών δημοκρατικών εξωτερικοτήτων σε μεγάλο βαθμό οι εθνικές πολιτικές κοινότητες δεν μπορούν να ρυθμίσουν αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή οι εθνικές δημοκρατικές διαδικασίες δεν μπορούν να ελέγξουν αυτούς τους μηχανισμούς που επιδρούν στην πολιτική τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δεν έχει μπορέσει να το κάνει. Και αυτό ακριβώς είναι η δεύτερη δημοκρατική της λειτουργία που ε, βρίσκεται στην ρίζα αυτής της κρίσης. Οπότε είτε θεωρούμε την κρίση ένα πρόβλημα στο συνηθισμένο πλαίσιο, δηλαδή ένα πρόβλημα της κοινωνικής ανευθυνότητας κάποιων κρατών ή ένα πρόβλημα χρηματοοικονομικών ροών και συναλλαγών, όπως και να το δούμε, έχουμε ένα δημοκρατικό πρόβλημα ή αδυναμία να ελεγχθούν οι διασυνοριακές αυτές ροές και η αδυναμία των εθνικών πολιτικών διαδικασιών να εσωτερικεύσουν το κόστος το οποίο επιβάλλουν σε άλλους. Αυτό σημαίνει και με την νομισματική ένωση, αλλά και σε άλλους τομείς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήδη. Η αδυναμία, η δυσκολία, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης είναι, κατά την άποψή μου, απλά συνέχεια της ε, δημοκρατικής αυτής αδυναμίας να εσωτερικευτούν οι εξωτερικότητες της αλληλεπίδρασης. Ως αποτέλεσμα λοιπόν του πολιτικού κενού που εμφανίζεται στην Ευρώπη, μεταξύ δηλαδή του επίπεδου και του εύρους των προβλημάτων και του επίπεδου και του εύρους της πολιτικής. Δηλαδή κάποια προβλήματα μπορούν να ρυθμιστούν αποτελεσματικά μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά η λύση οφείλεται στο ότι επειδή οι εθνικοί πολιτικοί χώροι δεν έχουν εσωτερικεύσει τα προβλήματα αυτά, δεν προμηθεύουν και τις λύσεις που πρέπει να υπάρξουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έλεγα πως το χάσμα αυτό είναι το σημαντικότερο δημοκρατικό έλλειμμα. Αυτό είναι, θα έλεγα, το θεμελιώδες ε, ζήτημα και οπωσδήποτε το ότι δεν έχει εσωτερικευτεί ακριβώς αυτή η αλληλεπίδραση οφείλεται στην έλλειψη αλληλεγγύης. Εγώ θα έλεγα πως η έλλειψη αλληλεγγύης αντί να είναι ζήτημα απουσίας πολιτικής ε, ή κοινωνικής ή οποιασδήποτε άλλης ταυτότητας είναι προϊόν της ίδιας αδυναμίας να εσωτερικευτεί η αλληλεπίδραση. Στην περίπτωση αυτή τα ωφέλη αυτής της αλληλεπίδρασης γιατί τα ωφέλη της αλληλεπίδρασης δεν έχουν ε, εσωτερικιστεί και άρα δεν μπορούμε να ε, επιδείξουμε την αλληλεγγύη που ε, απαιτείται. Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης που πρέπει να αναπτυχθούν πρέπει να πληρούν τους εξής όρους. Πρώτον, χρειαζόμαστε βεβαιότητα. Γι' αυτό κατά την άποψή μου απαιτεί μια σαφή πολιτική εξουσία. Δηλαδή η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να είναι τόσο διαχειμένη όσο είναι αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τους κινδύνους χρεοκοπίας κρατών στην Ευρώπη. Είναι σαφές πως αυτό δεν είναι δυνατόν στην Αμερική γιατί υπάρχει μια σαφής πολιτική εξουσία μπορεί να χρεοκοπήσει ε, δεν μπορεί να χρεοκοπήσει μια πολιτεία γιατί θα παρέμβει το ομοσπονδιακό κράτο. Αυτή η πολιτική δεν υπάρχει και κάτι σαν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα στην Ευρώπη. Το δεύτερο είναι πω πρέπει να αποκατασταθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη η οποία έχει πληγεί με την κρίση και κατά τη διάρκεια τη κρίση μεταξύ κρατών μελών και πολιτών στην Ευρώπη. Δεύτερον, χρειάζεται να καταστήσουμε σαφή και τα ωφέλη και τις δημοκρατικές συνέπειες της ε, αλληλεξάρτησης αυτής και θα κάνω κάποιες προτάσεις. Ε, τέταρτον, πρέπει να νομοποιήσουμε την δημοσιονομική αλληλεγγύη και αυτό θα γίνει, κατά την άποψή μου, μόνο εάν την εξηγήσουμε παράλληλα με τον πλούτο που δημιουργεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αυτό θα το τονίσω αργότερα. Πέμπτον, πρέπει να συνδέσουμε την πολιτική ενοποίηση με την οικονομική αλληλεγγύη. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει φορολογία χωρίς εκπροσώπηση και πως αυτή η εκπροσώπηση δεν σημαίνει κυρίως ε, θεσμικά όργανα, σημαίνει πολιτική. Δηλαδή, εάν έχουμε οικονομική αλληλεγγύη και μεταφορά κονδυλίων χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο και εκπροσώπηση ε, που θα θεωρείται θεμητή στα μαθήματα πολιτών, αλλά και το αντίστροφο. Δεν υπάρχει εκπροσώπηση χωρίς φορολογία. Δεν θεωρώ πως μπορούμε να αναπτύξουμε ισχυρή πολιτική εξουσία στην Ευρώπη χωρίς ε, κάποιο είδους αναδιανεμητική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω καμία πολιτεία η οποία μπορεί να επιβιώσει μέσω μακροπρόθεσμα εάν δεν βασίζεται σε κάποιο είδους αναδιανεμητική δικαιοσύνη. Οι πέντε αυτοί όροι έχουν αρχίσει σε έναν βαθμό να γίνονται αποδεκτοί και νομίζω πως ε, θα αποτελέσουν αντικείμενο συνέντηση, αν και ο βαθμός βεβαίως υλοποίησης τους είναι αντικείμενο συζήτηση γι' αυτό. ακούμε εκκλήσεις για μια δημοσιονομική ένωση. Αλλά τι εννοούμε ακριβώς. Αυτό είναι σαφές. Και Έχω ακούσει πολλούς και διάφορους να μιλάνε για δημοσιονομική ένωση και ε, νομίζω πως εννοούν διαφορετικά πράγματα. Νομίζω πως υπάρχουν τρία διαφορετικά πράγματα που είναι τμήμα της. Το ένα είναι έλεγχος των εθνικών διαδικασιών του προϋπολογισμού. Και βεβαίως υπάρχουν μετά στοιχεία δημοσιονομικής αλληλεγγύης, αν και αυτό το είναι πιο επίμαχο από το πρώτο και βέβαια υπάρχει το ζήτημα του ποιος είναι ο βασικός μηχανισμός, ο σωστός μηχανισμός. Και βεβαίως του πότε πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Και τρίτον, υπάρχει το στοιχείο της ανάγκης δημοκρατικής νομοποίησης και των νέων εξουσιών που θα πρέπει να αποκτήσει η Ένωση για να ελέγξει εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές και για να νομοποιήσει επίσης την ε, οικονομική αυτή και φορολογική αλληλεγγύη που θα πρέπει να προκύψει εντός της Ένωσης. Αυτά θα έλεγα είναι συνενετικά ε, όσον αφορά τις απαιτήσει της ε, ε, δημοσιονομικής αυτής Ένωση, αλλά τα μοντέλα είναι διαφορετικά. Θα προσπαθήσω να αναφέρω τρία πιθανά μοντέλα που προκύπτουν και προκύπτουν από τις ε, πρόσφατες ε, εξελίξεις στην Ευρώπη. Το ένα είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε μια ομοσπονδία κανόνων. Δηλαδή, θα αυξηθεί η εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εθνικές πολιτικές ε, του προϋπολογισμού, αλλά μέσω κανόνων, μέσω πειθαρχία. Η θέση εδώ πέρα, και αυτό ακριβώς προστάθηκε η συνθήκη με το νέο σύμφωνο σταθερότητας κτλ, πως ε, το πρόβλημα με το προηγούμενο σύστημα ήταν πως ε, οι κανόνες με το προηγούμενο σύστημα δεν ήταν οι σωστοί, δεν ήταν σωστή η επιβολή κτλ. Οπότε αν το αναπτύξουμε αυτό θα λειτουργήσει τελικά το σύστημα. Κατά την άποψή μου η πειθαρχία και οι κανόνες από μόνοι τους δεν θα δουλέψουν. Δεν θα δουλέψουν οικονομικά αν και δεν θα εστιάσω σε αυτό γιατί δεν ξέρω καμία νομισματική ένωση όπου ταυτόχρονα όλα τα κράτη είναι πλέον ασματικά. Δεν μπορούμε να έχουμε άρα μία ένωση χωρίς μηχανισμούς αναδιανομής. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να γίνει, να γίνει αυτή η αναδρομή. Αλλά και πιο σημαντικό, δεν θα λειτουργήσει πολιτικά. Θα υπονομεύσει την πολιτική και κοινωνική νομοποίηση της Ένωσης. Και αυτό γιατί είτε οι εθνικές πολιτικές ε, διαδικασίες θα διατηρήσουν μια αυτονομία οπότε θα αμφισβητηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των κανόνων ή η υποταγή τους σε ε, κάτι το μη πολιτικό, όπως θεωρείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αμφισβητήσει την ίδια τη δημοκρατία. Μία ένωση η οποία λειτουργεί μόνο με μαστίγια δεν θα ε, είναι κοινωνικά αποδεκτή από τους πολίτες ε, μέσω μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό νομίζω πως ως έναν βαθμό υπάρχει μία συνένεση πως το μοντέλο αυτό πρέπει να συνδεθεί με κάποια μορφή ε, δημοσιονομικής αλληλεγγύης και το μοντέλο άρα που υπάρχει εδώ πέρα ε, που εμφανίζεται ε, είναι σε κάποια στοιχεία της έκθεσης που είναι αν θέλετε μία ομοσπονδία εθνικών πολιτικών. Η πρώτη διάσταση η οποία υπήρχε και στο προηγούμενο υπόδειγμα είναι η μεταφορά των δημοσιονομικών εξουσιών στην Ένωση. Δεύτερον, κάποιος βαθμός αμοιβεοποίησης ή αν θέλετε αμοιβαία εξασφάλισης μεταξύ των κρατών μελών. Και το τρίτο στοιχείο, με το να υπάρχει η αμοιβαία εξασφάλιση της ε, χρηματοπιστωτικής ε, αλληλεγγύης. Το τρίτο σημείο που αφορά την νομιμοποίηση είναι ότι η νομοποίηση θα γίνεται κυρίως μέσα από τις εθνικές από τις εθνικές δημοκρατικές εξουσίες με μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και με μεγαλύτερη συμμετοχή στα τεκτενόμενα του Συμβουλίου. Αυτό φαίνεται να είναι ένα ανάμειγμα μεταξύ διακρατικής και ενωσιακής πολιτικής, αλλά εδώ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο τις πολιτικές Ευρωπαϊκές Ένωσης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος της, ε, των αποφάσεων που λαμβάνονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα παράδοξο. Βλέπουμε από τη μια μεριά ότι χάνεται η εξουσία της Κομισιόν. Η Κομισιόν μονάχα θέτει την πολιτική ε, ατζέντα, αλλά συγχρόνως έχει και ένα ρόλο ως εκτελεστής πολιτικών και ως ε, επόπτης της εφαρμογής της πολιτικής. Κατά την άποψή μου όμως αυτή η κατάσταση ουσιαστικά δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό χάσμα. Τελικά με τον τρόπο αυτό όλο και περισσότερο υποσκάπτεται η κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ένας από τους θεμελιώδεις λόγους για τους οποίους εγώ πιστεύω ότι το τωρινό μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν θα λειτουργήσει στον οικονομικό χώρο γιατί δίνει αρκετή πολιτική εξουσία. Θα είναι διάχυτη αυτή η πολιτική εξουσία. Θα εξαρτάται πάντα από τους εθνικούς πολιτικούς χώρους. Θα λειτουργεί μόνο με αυτόν τον τρόπο η οικονομική εξουσία με το τωρινό μοντέλο. Επίσης, θα πληγεί από ένα πολύ σοβαρό πολιτικό πρόβλημα και γιατί η δημοσιονομική αλληλεγγύη βασίζεται στις μεταφορές μεταξύ εθνικών κρατών και κάποιοι από τους πολίτες των χωρών που δίνουν τα χρήματα αυτά θα το βρίσκουν δύσκολο να αποδεχτούν μια τέτοια πολιτική και άλλοι οι οποίοι είναι αποδέκτες θα θεωρούν ότι υπόκειται σε μια πειθαρχία που θεσπίζουν άλλες χώρες. Θα υπάρχει λοιπόν η εξάρτηση όχι από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο αλλά από άλλα κράτη-μέλη. Και όπως σας λέω το βασικό πρόβλημα που έχουμε και που βρίσκεται στην πηγή της κρίσης είναι η αδυναμία να ενσωματώσουμε τους εθνικούς πολιτικούς χώρους σε ένα σύστημα αλληλεξάρτησης που πρέπει να διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιοδήποτε υπόδειγμα λοιπόν το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στους εθνικούς πολιτικούς χώρους θα αποτύχει. Αυτό είναι μία από τις κύριες παρατηρήσεις που θέλω να σας υποβάλω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα και να πάρουμε μέτρα για να ευρωπαϊκοποιήσουμε τους εθνικούς πολιτικούς χώρους. Γίνεται αυτό σε κάποια από τα άρθρα που σας έχω διανύμει βλέπετε ότι υπάρχει κάποια σειρά προτάσεων κάπως να υπάρχει δυνατότητα να γίνεται και μία ε, παρουσίαση της κατάστασης της Ευρώπης στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά δεν θα προχωρήσω για τα θέματα αυτά, γιατί πιστεύω ότι το μοντέλο αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα και έρχομαι σε ένα τρίτο μοντέλο το οποίο θα σας παρουσιάσω. Ένα πραγματικό υπόδειγμα δημοσιονομικής ένωσης αλλά με περιορισμένες εξουσίες, με τέσσερα κύρια στοιχεία σε αυτό το μοντέλο. και θα εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο το οποίο πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πιο βιώσιμο, όσο και δύσκολο να φαίνεται καταρχήν. Τα εξή τέσσερα στοιχεία περιέχει αυτό το μοντέλο. Ένα πραγματικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, νέε δομέ για τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζονται στο νέο δημιουργούμενο πλούτο και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου. Από τη δική μου πλευρά μόνο ένας πραγματικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να διορθώσει τα συμμετρικά σοκ της νομισματικής ένωσης και να δώσει και την απαραίτητη πολιτική εξουσία για μια νομισματική ένωση. Έχουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ που είναι το καλύτερο αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν δημιουργήθηκε η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, κάποιες από τις πρώτες μελέτες είχαν πει ότι τότε ήδη θα έπρεπε να είναι 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο προϋπολογισμός, ο κοινό προϋπολογισμός και έχει παραμείνει στο 1%. Κάποιες από τις βασικές λοιπόν προϋποθέσεις της Νομισματικής Ένωσης δεν έχουν υλοποιηθεί και αυτό μπορεί να εξηγεί εν μέρει την κρίση. Δεν θα πω τώρα στις λεπτομέρειες γιατί ένας προπολογισμό, είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς τους ασυμμετρικούς κλειδονισμούς. Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως των διαφθορτικών πολιτικών της. Πιστεύω ότι η μορφή και η φύση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνδέεται περισσότερο με τις εθνικές μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αναδιοργανώσει και να αναμορφώσει τις πολιτικές της ώστε να έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να προωθούν συστημικές αλλαγές στα κράτη-μέλη. Να το κάνω λίγο πιο απτό. Σκεφτείτε τα θέματα του, της έρευνας. Ένα από του τομείς όπου δαπανά πολλά χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει απλώς στα κράτη-μέλη, τις εθνικές αρχές, εθνικά σχέδια, χρήματα για να χρηματοδοτήσουν ερευνητικά προγράμματα, επί τη βάση των θεμάτων και των στόχων των εθνικών προγραμμάτων, τα χρήματα αυτά πρέπει να διαρθωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν σε μια συστημική αλλαγή στα ερευνητικά συστήματα των κρατών μέλων. Όχι να σας πούμε θα κάνετε, σας δίνουμε λεφτά για να κάνετε μελέτες στον α, β τρόπο, σας δίνουμε χρήματα για να κάνετε έρευνες σε ιδρύματα που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα των φοιτητών τους, των διδασκών τους, έχουν, ικανοποιούν κάποια κριτήρια αριστείας. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να έχει ένα πολύ πιο σημαντικό αντίκτυπο για να προωθήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Τέτοιου είδους συστημική, συστημικός αντίκτυπος θα γίνει και πιο ορατός για τους πολίτες. Η βασική ιδέα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει ένα ρόλο για την αναμόρφωση των κρατών μελών της, όχι μόνο μέσω του μαστιγίου, αλλά και μέσω της παροχής κινήτρων. Και ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται κίνητρα είναι με τη βοήθειά της να αναδιαθώσει τις πολιτικές στα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο αποτελεσματική σε εθνικό επίπεδο και πιο αποδεκτή συγχρόνως. Μια τρίτη πτυχή έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνδέονται με τις ευρωπαϊκές δράσεις και τον πλούτο που δημιουργούν. Το επιχείρημά μου είναι ότι η δημοσιονομική αλληλεγγύη θα γίνει μονάχα θεμητή στα μάτια των πολιτών όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδιανέμει τον πλούτο τον οποίο δημιουργεί η ίδια και όχι τον πλούτο κάποιων κρατών μελών. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα είναι απαραίτητο τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδέονται με δύο μορφές δράσης. Είτε η οικονομική δραστηριότητα η οποία γίνεται γιατί υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν κάνουμε μία μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και ένα τμήμα από αυτού, παραδείγματος χάρη το ΦΠΑ το οποίο είναι διαμεθοριακό να είναι ένα είδος φόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πόρος, αλλά δεν έχει τη μορφή φόρου για υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν αναπτύξουμε κάποιο τρίπο φορολογίας των πωλήσεων στο διαδίκτυο που είναι ένα, ήδη ένα τομέα όπου υπάρχει μεγάλο φορολογικό ανταγωνισμό, αν μπορούμε να αναπτύξουμε φορολογία στα θέματα αυτά, τότε οι πολίτε θα κατανοήσουν γιατί η Ευρώπη έχει αυτά τα χρήματα, είτε γιατί αυτή η δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που γίνεται δυνατή μόνο χάρη στην ύπαρξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικέ λοιπόν ε, δραστηριότητες και συναλλαγές υπάρχουν γιατί υπάρχει η εσωτερική αγορά, γιατί λοιπόν να μην παίρνει ένα τμήμα αυτού του κέρδους η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε γιατί υπάρχουν άλλοι τομείς όπου η φορολογική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε μια δράση που ελέγχει τις εξωτερικότητες μεταξύ των κρατών μελών. Παραδείγματο χάρη ένας φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένα φόρος στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, αλλά και ο φόρος για τις διαδικτυακές πωλήσει μπορεί να είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Μια τέτοια σχέση λοιπόν πρέπει να γίνει αυτή για του πολιτέ. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ο στόχος δεν είναι να δώσουμε <clears throat> απλώς περαιτέρω έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαν ένας πιο σημαντικός ρόλος είναι ότι από τη δική μου άποψη τα έσοδα και ο τρόπος με τον οποίο διαθρώνονται παίζουν θεμελιώδη χώρο, θεμελιώδη ρόλο για να κάνουν ορατό, ορατή στους πολίτες τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παρεχόμενη προσθέμενη αξία από την ύπαρξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα διαθρώσουμε τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο να κάνει ορατή για τους πολίτες την προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο δεν σημαίνει αυτή τη στιγμή, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. <clears throat> ένα τελικό στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι η ανάδυση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής σφαίρας. <clears throat> είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η πολιτική προβληματική για την ευρωπαϊκή πολιτική, για την ευρωπαϊκή πολιτεία ως, ως πολιτεία και όχι μονάχα η πολιτική υπέρ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο παρατηρήσεις. Το Κοινοβούλιο ή ένα μεγάλο μέρος του Κοινοβουλίου μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια κατεύθυνση. Πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υποστηρίξει ήδη την θετική του στάση εναντί μιας τέτοιας κατεύθυνσης. Εγώ αγωνίζομαι για το θέμα αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Ο Σάιμον Χίξ, ένας γνωστός πολιτικός επιστήμονας, έχει γράψει για τα θέματα αυτά. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οι εκλογές στην, ε, στο, του Ευρωκοινοβουλίου για ένα τρόπο επιλογής του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια τέτοια πολιτική αντιπαράθεση είναι απαραίτητη για να προωθήσει την ανάδυση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου και είναι σημαντική για να εσωτερικοποιηθούν οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ κρατών μελών που έχουν δημιουργηθεί με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το πλεονέκτημα εδώ είναι ότι αν οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γίνονται ένα είδος διελκυνστήνδος για την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να έχουμε διαφορετικές προτάσεις από τα πολιτικά ε, κόμματα, αυτό είναι διαφορετικό από μία πρόταση για την άμεση εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν και χωρίς καμία τροποποίηση των συνδικών. Αν τα πολιτικά κόμματα παρουσιάσουν αντιμαχόμενους υποψηφίους, καταρχήν οι ευρωεκλογέ θα έχουν να κάνουν με την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για τα πολιτικά προγράμματα των επικεφαλής της Κομισιόν. Ας υποθέσουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Η εξουσία λοιπόν και το κύρος που θα έχει ο τωρινός, θα έχει ο πρόεδρος της Κομισιόν για να υποστηρίξει τις προτάσεις του θα ήταν τελείως διαφορετικό αν αυτές οι προτάσεις είχαν επικυρωθεί με την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχαν επικυρωθεί και από μια ε, εκλογική πλειοψηφία που υποστήριξε αυτόν τον πρόεδρο στις εκλογές. Ένα βασικό στοιχείο λοιπόν θα είναι ότι όχι μονάχα θα ευρωπαϊκοποιήσουμε πλήρως τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό θα δώσει ένα πολιτικό κεφάλαιο, μια πολιτική αξιοπιστία και κύρο στον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι του Συμβουλίου. Γιατί αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία υποσκάπτουν το ρόλο τη Κομισιόν ω πολιτικού παίκτη και όχι ω τεχνοκρατικού μονάχα Και φυσικά αυτό θα δώσει στην Κομισιόν πολύ μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση. Και πιστεύω ότι το γεγονός ότι το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο προτείνει στο Κοινοβούλιο τον πρόεδρο της Κομισιόν κάνει οτιδήποτε. Είναι σαν τα προεδρικά συστήματα που έχουν πολλές χώρες όπου ο πρόεδρος πρέπει να διορίσει τον Πρωθυπουργό αλλά λαμβάνοντας υπόψη τους τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτό δεν αλλάζει καθόλου τα ουσιαστικά, τον ουσιαστικό τρόπο διορισμού του Πρόεδρου της Κομισιόν. Και θα κλείσω λοιπόν με αυτό γιατί νομίζω ότι έχω ήδη χρόνο τριβήσει και έχω μακρηγορήσει. Αν λοιπόν προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή θα υπάρχουν και ελοχεύοντες κίνδυνοι. Φυσικά άμα πολιτικοποιήσουμε την εκλογή του Πρόεδρου της Κομισιόν και είμαι εν επιγνώση αυτών των κίνδυνων, αλλά νομίζω τα δυνητικά ωφέλη ξεπερνούν τους κινδύνους και θα παραμείνει βέβαια και κάποιο στοιχείο ότι θα είναι κατά κάποιο τρόπο πολύμορφη η Κομισιόν γιατί οι εθνικές κυβερνήσεις θα υποστηρίζουν διαφορετικές απόψεις και επομένω και η σύνθεση της Κομισιόν θα είναι ακόμα πολύ μορφή από ιδεολογική έποψη. Από την άλλη μεριά όμω. αυτό θα μειώσει, θα μειωθεί πρώτον γιατί ο πρόεδρος της Κομισιόν ως αυτός ο οποίος επελέγει από τις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου θα έχει και το κύρος έναντι των εθνικών ε, κυβερνήσεων για την επιλογή των μελών της Κομισιόν θα έχει πολύ καλύτερη διαπραγματευτική θέση στα θέματα αυτά και θα έχει και μεγαλύτερο κύρος ο ίδιος μέσα στην Κομισιόν. Η δική μου προσδοκία είναι ότι αν το σύστημα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή και σας λέω ότι αυτό δεν, απαιτεί μια συνταγματική τροποποίηση στις συνθήκες, μπορεί να προκύψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που ονομάζω ένα διαφορετικό είδος ημιπροεδρικού καθεστώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Κομισιόν είναι το εκτελεστικό σώμα και ο κύριος πολιτικός ε, παίκτη που έχει ένα ηγετικό ρόλο, που θα εξαρτάται και θα υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο και θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την άλλη πλευρά το Συμβούλιο θα παίζει το ρόλο αυτού που έχει το δικαίωμα αρνησή κυρίας, όπως ένα προεδρικό σύστημα. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να εξελιχθεί το σύστημα. Αν δεν κινηθεί το σύστημα προς την κατεύθυνση αυτή, ο κίνδυνος είναι αυτός που βλέπουμε σήμερα, ότι θα υπάρξει μια αύξηση στο ρόλο του Συμβουλίου και το Συμβουλίο θα γίνει ο κύριος και ο μόνος σχεδόν πολιτικός παίκτη. Για τους λόγους λοιπόν που ανέφερα στην αρχή της παρουσίασής μου, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή, που είναι ένα πρόβλημα πολιτικής φύσεως, είναι ότι αν δεν υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη προς το σύστημα που ανέφερα, τα αποτελέσματα θα είναι κυρίως αρνητικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον καθηγητή Μαντούρο. Λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να εγκαταλείψω την Προεδρία. Θα με αντικαταστήσει ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Λυπάμαι που δεν θα ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και ακόμα περισσότερο τις δικές σας απαντήσεις. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ θα έρθει εδώ. Και ο πρώτος που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο κ. Σέφλινγκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον καθηγητή Μαντούρο για μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω και εγώ ορισμένε σκέψεις οι οποίες δεν νομίζω ότι είναι αντίθετες με αυτά τα οποία είπατε αλλά ίσως να διευρύνουν Γνωρίζω και εγώ το Σάιμον Χίξ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αναφερθήκατε καταρχάς It seems to me that this is absolutely right. I mean, I agree with the democratic failure proposition. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να συνδέσουμε. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι τα κράτη-μέλη μεταξύ τους ουσιαστικά έχουν προχωρήσει, προχωρήσει στην αποσύνδεση των διαφόρων επιπέδων, όχι ανάμεσα στη μία τα κράτη-μέλη και στην άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μεταξύ τους. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά αναπτυσσόμενη ανάμεσα στο βορρά και στο νότο, πάντα υπήρχε βέβαια κατά κάποιο τρόπο και μια αντίστοιχη διαφοροποίηση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή και αυτό επηρεάζει το επίπεδο των μεταρρυθμίσεων που προτείνεται. Δεν είμαι βέβαιος για το ότι μέχρι ότου αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σας θα μπορούσαν, να μπορούσαν να καρποφορήσουν. Δεύτερον, μιλήσατε για την εσωτερήκευση. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείτε. Εγώ έχω μια αντίληψη για τη λέξη αυτή η εσωτερικευσή, αλλά δεν είμαι βέβαιος αν συμφωνούμε. Εάν πράγματι αυτό το οποίο λέτε είναι να προχωρήσουμε στη συνειδητοποίηση την καλύτερη της ευρωπαϊκής διαδικασίας, το θέμα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και αν μπορούμε να το κάνουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή σας. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για τον χρονισμό και κατά πόσον συνειδητοποιείται την κρισιμότητά του. Γιατί από τη μία υπάρχουν ε, ε, διαφορετικά συμφέροντα πολιτικά και οικονομικά, μας ε, τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις και το θέμα είναι πώς θα τα ενσωματώσουμε όλα αυτά, πώς θα τα εσωτερικεύσουμε όλα αυτά στο σωστό χρόνο. Σχετικά με την αναδιαμητική δικαιοσύνη θα έλεγα αυτό είναι πολύ σωστό. Να προσθέσω μια μια κοινωνιολογική διάσταση. Εγώ ήμουν πολιτιολόγος, αλλά ενδιαφέρομαι ακόμα και σήμερα σαν πολιτικός για τις κοινωνικές διαδικασίες. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια δημογραφική θα έλεγα παρακμή που δημιουργεί μια θα έλεγα δημογραφική ανασφάλεια και και αυτό δημιουργεί μια οικονομική ασφάλεια για τις γενεακές σχέσεις, διαγενειακές σχέσεις και βάζει σε δεύτερο επίπεδο θα έλεγα τις ε, προσπάθειες κάλυψης αναγκών των άλλων νότιων, ανατολικών και, τα λοιπά. Φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδος των βαλτικών χωρών, των βασικών έξι, μαζί με τη Φιλανδία τη Φιλανδία και τη Δανία. Αυτός είναι ένας άλλος πόλος αν θέλετε, είναι μια άλλη μορφή διάφρωσης των αναπτυσσόμενων διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο καθιστά τις προτάσεις σας λιγότερο εύκολο να εφαρμοστούν, εύκολες στην εφαρμογή τους. Για την αναδιανομή πάντως της, σε εισαγωγικά δικαιοσύνης είναι κάτι το οποίο συμφωνώ. Μιλήσατε για την δημιουργία ενός πολιτικού χώρου. Εγώ το ονομάζω αυτό δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εισαγωγικά πόλεως με την αρχαία έννοια. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχουμε αυτό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια πολύ μεγαλύτερη παρουσία στα κράτη-μέλη από τη σήμερα. Αναφερθήκατε στα θέματα της φορολογίας. Συμφωνώ όχι για λόγους εισοδήματος, αλλά με στόχο την δυνατότητα της μεγαλύτερης εμπλοκής των πολιτών. Και έχετε δίκιο. Θα το πετύχουμε αυτό αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θα έλεγα παρούσα σε εισαγωγικά στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή μαζί της άμεσα οι πολίτες. Δεν θα συμβεί αυτό από τη μια μέρα στην άλλη βέβαια, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ και ένα θέμα συνέπειες θα έλεγα, οι διαφορετικές μορφές εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων. Ε, οι πολιτισμοί εφαρμοστικοί είναι διαφορετικοί πολύ μεταξύ τους. Πολλοί από τις εκλογέ μου στην Ουγγαρία μου λέγουν γιατί εμείς στην Ουγγαρία κάνουμε αυτό, ενώ στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες κάνουν κάτι το εντελώς διαφορετικό. Αυτό λοιπόν έχει άμεση σχέση με το θέμα της αλληλοεξάρτησης, την οποία όλοι βιώνουμε, αλλά οι διαφοροποιήσεις αυτές δημιουργούν προβλήματα και πολλές φορές κάποιες δυσάρεστες πολιτικές οι κυβερνήσεις των κρατών μελών τις εφαρμόζουν λέγοντας ότι είναι κοινοτικές πολιτικές και αυτό δεν βοηθάει. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια εποπτική αρχή Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να διασφαλίζει την ταυτόσιμη εφαρμογή των κοινοτικών ρυθμίσεων. Έτσι θα μπορέσουμε να νομιμοποιήσουμε την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ανάγκη και για μια πιο συμβολική διάσταση και νομίζω ότι απαιτείται άμεσα να ενισχυθεί η κοινοτική παρουσία. Ε, μια φράση ακόμα. Ένα στοιχείο επιπλέον και θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Είναι ο λόγος ο τεχνικός και ο νομικός τον οποίο χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να μετατραπεί σε πολιτικό λόγο για να γίνει κατανοητός. Ο κύριος Ραντζέλ. Έχουμε μέχρι τις 12.45. Αλλά ξέρω ότι είναι πολλοί αγορητές. Σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να χαιρετήσω τον καθηγητή Μαντούρου. δεν είναι μονάχα ένας λαμπρός Πορτογάλος και Ευρωπαίος ερευνητής και διανοητής, αλλά και πολύ καλός φίλος. Όταν προσπάθησα να κάνω κάποια έρευνα, πήγα στη Γαλλία κάποιους μήνες και ζούσα στο σπίτι του και καθηγητή Μαδούρου. στη Φλωρεντία, συγγνώμη, όχι στο Παρίσι, ζούσα στο σπίτι του. Και έχει μια άλλη αρετή ο κύριος Μαντούρου. Πάντα προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την ε, φιλία μας με τον Βιτάλ Μορέιρο Και όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ καλές αναμνήσεις που έχω Όλα αυτά δείχνουν την πολύ σημαντική συμβολή που έχει κάνει ο κ. Μαντούρο για να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό πολιτικό χώρο. Έρχομαι τώρα. Θα συνεχίσω στα πορτογαλικά. Θέλω να χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτή την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να σχολιάσω <clears throat> σε σχέση με αυτά που είπε ο Μαδούρο είναι δύο ή τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη διάγνωση την οποία μας παρουσίασε. Και δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει μονάχα για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη είναι μια περίπτωση η οποία είναι αποκαλυπτική και εμβληματική για αυτά τα προβλήματα. Έχουμε το θέμα της αποεδαφικοποίησης της εξουσίας υπάρχει μια διάχυση και μια διαφοροποίηση μεταξύ αυτού που ήταν το παλιό ε, μοντέλο της εξουσίας που βασιζόταν σε εκλογικές περιφέρειες. Βρισκόμαστε λοιπόν όλοι σε εκλογικές περιφέρειες οι οποίες όμως δεν έχουν την εξουσία. Η εξουσία βρίσκεται αλλού. Οι βασικέ αποφάσει παίρνονται αλλού. Εμεί, παραδείγματο στην Πορτογαλία, ξέρουμε ότι οι βασικέ αποφάσει λαμβάνονται κάπου αλλού. Παραδείγματο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχει πραγματικά αυτό το χάσμα, αυτή η απόκληση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι όχι μόνο ευρωπαϊκό, είναι ένα παγκόσμιο. Στην Ευρώπη είναι πιο έντονο ακόμα γιατί υπάρχει και αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τη διάγνωσή σας. Θα ήθελα να τονίσω επίσης όπως έχω ακούσει <clears throat> και από πάρα πολλούς να το λένε τα, τα χρόνια αυτά της κρίσης και μετά από αυτά που είπε ο, αυτά που είπε ο Υπουργό τη Πολωνία Εξωτερικών και Οικονομικών κ. Σικόρσκι ήταν τα πιο ενδιαφέροντα. Γιατί τόνισε την ανάγκη να υπάρξει μια πολιτική και συνταγματική αντιμετώπιση. Και σας υπενθυμίζω αυτή τη φράση, ότι δεν αρκεί να υπάρχει να μην υπάρχει φορολογία χωρίς αντιπροσώπευση που ήταν το σύνθημα της Αμερικανικής ε, επανάστασης δεν πρέπει να υπάρχει και α, να αντιπροσώπευση χωρίς φορολογία. Και έρχομαι στο τρίτο μοντέλο της αλληλεγγύης που ανέφερε ο κ. Μαντούρο. Πού είναι τα δύο ερωτήματά μου. Καταρχήν η έννοια της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές συστημικής παρέμβασης οι οποίες θα εξασφαλίσουν αυτή την πολυεπίπεδη δημοκρατία. Από τη μία πλευρά έχουμε τα εθνικά κράτη και τα εθνικά κοινοβούλια φυσικά. Υπάρχει δηλαδή η εθνικοποίηση των πολιτικών και μπαίνουν όλο και περισσότερο οι εθνικοί φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Θεσμή και η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή προωθεί αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κίνηση και πάλι προς τα εθνικά κράτη της ευρωπαϊκής πορείας. Συγχρόνως όμως υπάρχει και η αντιθέτη τάση. Παραδείγματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε συστηματικά την εσωτερική κατάσταση διαφορών κρατών. Λέγουμε ότι γίνεται αυτό και εκείνο το α ή το β κράτος, όπως είδαμε με τη Ρουμανία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει η συστηματική παρουσία πολιτικών θεμάτων που αφορούν την εσωτερική κατάσταση των κρατών μελών δημιουργούν και μία προβληματική. Υπάρχουν, υπάρχει λοιπόν μια διάχυτη πολιτική σφαίρα η οποία δεν υπόκειται σε σαφείς κανόνες και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Για την τελική σας πρόταση εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρξει μια εκλογή του Πρόεδρου της Κομισιόν από τις ευρωεκλογικές. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε για το ημιπροεδρικό σύστημα και τον ρόλο που θα πρέπει να έχει το Συμβούλιο, ότι πρέπει κάπως να μειωθεί η υπερβολική εξουσία του Συμβουλίου. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι από συνταγματική έποψη το Συμβούλιο και ιδίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι η διάσκεψη κορφή των ηγετών έχει και κλείνω, έχει μια αμφισημία στη μορφή του δεν είναι ένα όργανο το οποίο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αλλά είναι αυτό το οποίο δίνει και κατευθύνσεις συγχρόνως. Έχει λοιπόν ένα έμεσο νομοθετικό ρόλο. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει... Αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό, το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου. Αυτό το όργανο το οποίο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις να έχει συγχρόνως και ένα είδος νομοθετικής εξουσίας. Ή λοιπόν θα δώσουμε νομοθετικό ρόλο στο Συμβούλιο και θα αφήσουμε την πολιτική εξουσία στην Κομισιόν ή αλλιώς θα πρέπει να πάβει το νομοθετικό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχει νομοθετική εξουσία και θα πρέπει αυτή η εξουσία να παραμείνει στις ειδικευμένε μορφές και σχηματισμούς του Συμβουλίου. Εδώ είναι λοιπόν η δική μου ε, αντίρρηση σε αυτή την τελευταία την πρόταση που θεωρείται ότι θα λύσει το πρόβλημα κύριε Μαντουρό. Κύριε Στασκόφσκι πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά τα οποία λέτε, αλλά έχω κάποιες πρακτικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ε, πραγματική δημοσιονομική ένωση είναι θαυμάσια ιδέα, αλλά όταν μιλάμε για την έκθεσή μας για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, ε, για ποιον, για 27 κρατημέλη, για όσους έχουν υπογράψει το δημοσιονομικό σύμφωνο ή για τους 17. Εάν είναι για λιγότερους από 27, τότε τι σχέσεις θα έχουμε μεταξύ αυτών που θα είναι μέσα και των έξω. Και μιλάτε για προπολογισμό της Ένωσης. Θα έχουμε δύο προπολογισμού, έναν για τους 27 και έναν πραγματική δημοσιονομική ένωση, γιατί αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Και όταν μιλάμε για το βαθμό πολιτικής βούλησης, το εάν τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα ήθελα να έχουν πραγματικά μια τέτοια ένωση 27. Κατόπιν προτείνεται μια επανάσταση και ξέρουμε πώς δουλεύει η ένωση. Αργές λήψεις αποφάσεων, παζάρια κτλ. Εάν είναι να αλλάξουμε... Εγώ συμφωνώ πλήρω με τις συνταγές σας, αλλά το να αλλάξει ο προπολογισμό να τριπλασιαστεί, να αλλάξει η δομή των πολιτικών της Ένωσης για να προωθήσουν την αλλαγή και να δημιουργηθεί ένας πολιτικός χώρος είναι πολύ ωραίο σενάριο. Το προσυπογράφω, αλλά το ερώτημα είναι εάν μπορεί να γίνει γρήγορα. Οι απαντήσεις που χρειαζόμαστε θα πρέπει να γίνουν γρήγορα και φαίνεται πως οι αποφάσεις αυτές θα χρειαστούν χρόνο για να εφαρμοστούν. Το ζήτημα μετά κατόπιν της νομοποίησης ε, γιατί αυτές οι ιδέες για τη δημιουργία ενός πολιτικού χώρου υπάρχουν, αλλά δυστυχώς θεωρώ πως πρώτα απ' όλα χρειάζεται ισχυρή νομοποίηση τώρα εάν για να προχωρήσουμε και θα χρειαστεί καιρός για τους πολίτες να ε, κάνουν κάτι τέτοιο. Ακόμα και αν ε, εισαχθεί παραδείγματο χάρη μια σύνδεση με τις ευρωεκλογέ και τις εκλογές του Πρόεδρου της Επιτροπής δεν θα το δουν οι πολίτες αυτόματα. Επίσης για φόρους μιλάτε. Και πάλι νομίζω πως συμφωνώ με τη φιλοσοφία σας, αλλά δεν θεωρώ πως εάν είναι να βάλετε ένα φόρο στις συναλλαγές του διαδικτύου, θα πούνε οι πολίτες «Α, να τα τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Όχι, περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσουμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Γιατί μόνο 8% των πολιτών κάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο με άλλη χώρα. Και ούτω ή άλλω δεν του αρέσει τους φόρους, ε, δεν αρέσει στον κόσμο, δεν αρέσει στον κόσμο οι φόροι. Και θα είναι τελείω αντιπαραγωγικό να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και τέλος, ε, η ερώτηση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλα αυτά. Γιατί μιλάτε για νομοποίηση και το τεράστιο αυτό κενό στην εσωτερήκευση των ωφελών κτλ. Πολλοί προτείνουν πως ε, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να παίζουν το ρόλο της νομιμοποίησης. Ή τι θα γίνει. Κάποιο μείγμα των δύο που μονίμως θα μας υποκαθιστούν τα εθνικά κοινοβούλια. Ποια είναι η αποψή σας λοιπόν για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προφανώς αυτό σχετίζεται και με το πρώτο ερώτημα, δηλαδή πραγματική δημοσιονομική ένωση για ποιον και θεσμικά πώς θα γίνει και θα μπω σε λεπτομέρειες σχέσεων μεταξύ του Συμβουλίου, Προέδρου του Συμβουλίου, της Κομισιόν κτλ. γιατί θα φάμε πολύ ώρα. Για εμένα τα σημαντικότερα ερωτήματα είναι αυτά τα οποία ανέφερα. Ευχαριστώ. Κύριε Μαντέρο, ελπίζω να τα σημειώσατε, γιατί Θα ακούσουμε όλες τις ε, ερωτήσεις και θα τις απαντήσετε μία και καλή στο τέλος. Έχουμε τέσσερις ακόμα ομιλητές και να έχετε κατά νου πως ε, όσο συντομότερε οι ερωτήσεις, τόσο καλύτερες και οι απαντήσει. Γιατί 12.45 θα τελειώσουμε. Έμα, αυτό εξαρτάται από εσά. Γιολάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά συναρπαστικό να είναι κανείς στην ΑΦΚΟ γιατί μπορεί να αναπτύξει την ε, σκέψη του. Γιατί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος μιλάει κανείς το πολύ για, για δύο λεπτά, αλλά εδώ πέρα μπορεί πραγματικά να αναπτύξει σκέψη του. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε κύριε Μαδούρο. Από τις τρεις παραλλαγές που προτείνατε, η τρίτη παραλλαγή νομίζω είναι αυτή η οποία θα προχωρήσει στο πλαίσιο των συνθήκων και μια παραλλαγή στην οποία έχουμε ήδη κάνει αρκετή προεργασία. Ένας πραγματικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με δικά μας έσοδα και υψηλότερος βεβαίως με 1% του ΑΕΠ δεν μπορούμε με 27-28 χώρες να βρούμε την ισορροπία. Το επόμενο είναι η ευρωπαιοποίηση, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, ξέρετε, η έκθεση DAF αναβλήθηκε για τρίτη φορά. Δηλαδή δεν καταφέρνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το φέρει αυτό στην Ολομέλεια. Αυτή είναι μια πραγματική αδυναμία. Δεν είμαστε σε θέση να περάσουμε με πλειοψηφία την έκθεση DAF. Βεβαίως, εντάξει, μπορούμε να έχουμε υποψηφίους ε, των κομμάτων χωρίς την έκθεση Αλλά το πρόβλημα είναι πως δεν έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουμε 27 εθνικές εκλογές και χωρίς μια ενιαία λίστα δεν έχουμε ευρωπαϊκά κόμματα. Χρειάζεται ένα στοιχείο, μια εντολή για τα ευρωπαϊκά κόμματα. Στα 11 αυτά πιστοποιημένα κόμματα και τότε θα έχουμε μια πραγματική διεθνή συζήτηση. Αλλά ε, δύο ερωτήσει και ο κύριος Στασκόφσκι έθεσε το ίδιο ερώτημα το εάν είναι όλα αυτά όνειρα. Γιατί δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο η Μεγάλη Βρετανία και κάποιοι άλλοι ίσως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Τι θα κάνουμε λοιπόν εάν δεν ε, συμμετάσχουν και οι 27. Μετά. Δημοσιονομική Ένωση σημαίνει και κοινή ανάληψη χρέους. Το αναφέρατε. Εκεί πέρα έχουμε πιθανώς συνθήκες με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν συμφωνεί κάτι τέτοιο με τη συνθήκη, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την συνθήκη ή πώς χρειαζόμαστε μια νέα συνθήκη για να γίνει κάτι τέτοιο ή υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κάτι εκτός της συνθήκης, ως μια διακυβερνητική συμφωνία. Εκεί πέρα βεβαίως δεν θα έχει ρόλο ούτε η Κομισιόν, ούτε το Κοινοβούλιο. Και τα εθνικά κοινοβούλια πιθανώς θα έχουν ένα ρόλο και θα έχουμε νέες δυσκολίες νομιμοποίησης. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, ευχαριστώ, κύριε και ο Γκολτιέρη. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Και συμφωνώ με την βασική θέση του ομιλητή Ο πυρήνας του προβλήματος είναι αυτό που είχε πει ο Γκράμψη, είναι η αντίθεση ανάμεσα στον κοσμοπολιτισμό της οικονομίας και τον εσωτερικό εθνικισμό της πολιτικής. Ακριβώς λοιπόν λόγω της πολιτικής φύσης τελικά του προβλήματος στα πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων και των εθνικών πολιτικών το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν προβλήματα βέβαια με το σύμφωνο σταθερότητας, Βέβαια οι επιπτώσεις στο εσωτερικό νομοθετικό πλαίσιο, οικονομικό συγγνώμη πλαίσιο, μπορεί να μετατραπεί και σε νομικό πρόβλημα το οποίο μερικές φορές είναι αξεπέραστο. Τώρα για την λεγόμενη φορολογική ένωση η οποία να πάνω στην έννοια των ιδίων πόρων, ισχυρών ιδίων πόρων, όπως έλεγε ο κύριος Μαντούρο, νομιμοποίηση και αναδιανομή Το πρόβλημα είναι ότι από τη μία ο Μαντούρο αυτό το οποίο ζητά είναι πιο ρεαλιστικό από ό,τι ζητούν άλλοι γιατί θα, μπορούσε αυτά τα οποία, θα μπορούσαν αυτά τα οποία είπε να εφαρμοστούν με τις ισχύουσες συνθήκες, όσοι έχουν τα πράγματα σήμερα από την άλλη όμως και ταυτόχρονα οι διαδικασίες τις οποίες ζητούν οι συνθήκες αντικειμενικά δεν είναι ιδιαίτερα ρεαλιστικές, γιατί αν απαιτείται ομοφωνία για τους νέους πόρους, αν πρέπει να υπάρξει ομοφωνία για τον καθορισμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα σπάσει το φαύλο κύκλο. Και δεν υπάρχει και επαρκής νομιμοποίηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να της δοθούν περισσότεροι πόροι και να μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει σωστά. Και ταυτόχρονα το θέμα της νομιμοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει σε εκκρεμότητα. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς θα μπορέσει κανείς να διανύσει αυτή τη διαδικασία με τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και με τους περιορισμούς τους διαδικαστικούς και θεσμικούς που υπάρχουν σήμερα. Γιατί δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο, ε, έχουμε δει πολλά θεωρητικά σενάρια. Μπαίνοντα λίγο στην ουσία του πράγματος, είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να ορίσει ακόμα και τεχνικά και διαδικαστικά τις ιδέες του κυρίου Μαντούρο σε ορισμένους τομείς. Τη διαδικασία για τους ιδίους πόρους, σαν παράδειγμα. Πώς μπορεί να συνδυάσει στο εσωτερικό του κοινοτικού πλαισίου και εδώ θα συμφωνήσω με τον Τσαρκόφσκι γιατί αυτό θα πρέπει να είναι βασικό χαρακτηριστικό της πρότασής μας. Να χρησιμοποιήσει κανείς διαφοροποιούμενες διαδικασίες όπως το άρθρο 136, την ενισχυμένη συνεργασία, την σύγκληση ανάμεσα σε κράτη-μέλη, πώς όλα αυτά να μπορέσουμε να τα εντάξουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα συνδέσουμε με το διοργανικό πλαίσιο, με τα τρία μεγάλα όργανα, γιατί εκτός αυτής της διοργανικής συνεργασίας δεν μπορεί να υπάρξει νομιμοποίηση πολιτική. Αυτό είναι το δίλημα λοιπόν για το οποίο πρέπει εμείς να κάνουμε κάποιες προτάσεις για λύση. Θα πρέπει φυσικά να υποδείξουμε κάποιο δρόμο, τον οποίο εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως τον προτείνεται είναι σωστός, πρέπει ταυτόχρονα να προτείνουμε και μια σταδιακή διαδικασία, η οποία με τον τρόπο να καθιστά την επιλογή του δρόμου αυτού ελκυστική και εφικτή φυσικά. Κάποιες από τις ιδέες σας όπως η σύνδεση του 136 με το 152 ε, ομοφωνία για το 17, ε, ανάμεσα στους 17 ταυτόχρονα λέγοντας ότι η ψηφοφορία για την Ευρωζώνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το οποίο είναι νομικά ισχύον. Λοιπόν, και τεχνικά οι προτάσεις του Μαντούρο νομίζω ότι είναι λοιπόν εφικτές. Επανήλθα, λέει ο κύριος Καθίνη. Λυπάμαι που δεν άκουσα την ομιλία του κύριου Γκουαλτιέρη. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Μπρόνς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλω να σταθώ στο τελευταίο σημείο. Λέτε ότι μπορούμε να πείσουμε τους εκλογείς να επιδεχθούν ευρωπαϊκά κριτήρια για τον τρόπο με τον οποίο θα ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές. Και χωρίς να είμαι πατερναλιστής, Προσθέτετε και τη σημασία, θεωρείτε ότι αν προσθέσετε τη σημασία της επιλογής του Πρόεδρου της Επιτροπής, αυτό θα ευρωπαϊκοποίηση εκλογέ. Αυτό γίνεται στι βουλευτικέ εκλογέ. Ξέρουν αυτοί που ψηφίζουν στι βουλευτικέ εκλογέ δεν ψηφίζουν μονάχα τον άμεσο εκπρόσωπό του, αλλά ότι εκλέγουν έμεσα και τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Αλλά μόνο και μόνο να το προσθέσουμε αυτό σε ευρωεκλογέ δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκλέγουν οι πολίτε. Και δεν μπορείτε τελικά να το επιβάλλετε ο κόσμος έχει το δικαίωμα όχι μόνο να ψηφίσει αλλά και να αποφασίζει τα κριτήρια από των οποίων βασίζεται η θέση του στις εκλογέ, όσο και αν στενοχωρεί πολλού αυτό. Νομίζω ότι οι αλλαγές στην πολιτική ταυτότητα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές, σε συνταγματικέ αλλαγές. Αλλά και το αντίθετο θα μπορούσε να γίνει. Αλλά στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι πολύ δελαστικό για τα κόμματα να χρησιμοποιούν την έλλειψη δημοφιλίας των αντιπάλων τους για να προσποριστούν κάποιο, α, κάποιο κέρδος. Θα πρέπει να είναι ένα πάρα πολύ πειθαρχημένο κόμμα που θα πετάξει αυτό το πλεονέκτημα και θα βασιστεί μονάχα στα ευρωπαϊκά θέματα. Οι δικές μας εκλογές, οι δικές μας ευρωεκλογές βασίζονται σε εθνικά κριτήρια. Ο ένας στους 100 ίσως σκέφτεται περισσότερο την Ευρώπη από ότι τα εθνικά προβλήματα και τις εθνικές αντιπαραθέσεις. Αν επανέλθουμε στο θέμα της αμοιβαιοποίησης του χρέους και των βαρών και των ωφελών του προπολογισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να το πετύχουν αυτό ή να το δεχτούν οι εκλογείς, πρέπει να υπάρχει μια κοινή ταυτότητα. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε μια χώρα δέχονται τα λεφτά που δίνουν σε να πηγαίνουν σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ίδιας χώρας τους. Αλλά όσο δεν υπάρχει μια κοινή ε, ταυτότητα, δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το αν θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα ή όχι <clears throat> μεταξύ μας. Αλλά απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το είδαμε αυτό με την ε, δυσφορία των Γερμανών εκλογών εκλογέων στην ιδέα ότι οι φόροι τους, τουλάχιστον έτσι το βλέπουν, χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν και να επιδοτήσουν την Νότια Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι κοινέ ταυτότητες θα πρέπει να προϋπάρχουν πριν αντιμετωπίσουμε τα θέματα της αμοιβαιοποίησης του, του χρέους και όχι να έπονται αυτή τη απόφαση για Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Χέφνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο για να υπάρξει χρόνο και για απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Είχε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και όσον αφορά την ανάλυση και τις προτάσεις. ήμασταν περισσότερο θα έλεγα στο επίπεδο των τίτλων και δεν μπορέσατε με λεπτομέρειες να μας πείτε πώς ε, τα βλέπετε τα πράγματα λεπτομέρως. Τόσο, έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά μία μόνο θα θέσω. Έχετε δίκιο, κατά την άποψή μου. Τα προβλήματα είναι ένα πρόβλημα δημοκρατίας και αυτό το οποίο θα ρωτούσα εγώ είναι τι σημαίνει αυτό για την διαδικασία. Δεν μιλάω για τις θεσμικές προτάσεις, αλλά για την διαδικασία της λύσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο με απασχολεί πολύ. Αυτή τη στιγμή ολόκληρη η Ευρώπη ε, αναρωτιέται το τι θα κάνουν οι τέσσερις ε, Μπαρόζο, Γιούνκερ, Φανρόμπο και Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται ως εξής πάντα όλο ένας μικρότερος αριθμός ανθρώπων έχει όλο και περισσότερη εξουσία. Και εμείς ε, ως κοινοβούλιο μπαίνουμε πλέον στον ρόλο του θεατή. Οπότε το ερώτημά μου είναι πώς μπορούμε την διαδικασία αυτή να την συμβιβάσουμε με τον δημοκρατικό έλεγχο και την νομοποίηση εντός της ε, μεθόδους. Πρέπει να, τη μεθόδου πρέπει να διαμορφωθεί αυτή η διαδικασία ώστε να υπάρχει και αποδοχή ε, και νομοποίηση και να δημιουργεί νομοποίηση όχι να καταναλώνει αν θέλετε. Ποιος θα μπορούσε να είναι λοιπόν ο ρόλος του Κοινοβουλίου εδώ πέρα. Δεν έχουμε κάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Όσοι ήθελαν το λόγο μπόρεσαν να μιλήσουν. Γι' αυτό θα πρέπει να απαντήσετε σε πέντε περίπου λεπτά. Δέκα λέει ο κύριος Γουαλτιέρη. Θα προσπαθήσω. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και τα σχόλια, αλλά θα, προσπαθήσω ξεκινώντας από αυτό το οποίο μου φαίνεται ένα κοινό κομμάτι όσον αφορά το αδύνατον του πράγματος, το πολιτικά αδύνατον όχι νομικά δυνατόν. Θα κάνω κάποια σχόλια, θα το αφήσω σας το πώς θα κάνετε. Εγώ είμαι πανεπιστημιακός. Νομίζω πως θα κανετε εγω ειμαι παρεπιστημιακος νομιζω πως βασικα τις προάλλες πρόσφατα έγινε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο με πολλούς πανεπιστημιακούς και ειδικού για την ευρωκρίση και το τι μπορούμε να κάνουμε και άκουσα τις διάφορες προτάσεις για αμοιβαιοποίηση του χρέους, ευρωμόλογα κτλ. Και μετά έκανα την πρότασή μου και άκουσα τις ίδιες δηλώσεις πως αυτό είναι αδύνατον. Και η απάντησή μου ήταν, μα επί δύο ημέρες συζητάμε τις αδύνατες προτάσεις της δικές σας, γιατί να μην συζητήσουμε και τη δική μου αδύνατη πρόταση. Γιατί στην πραγματικότητα οποιαδήποτε άλλη πρόταση είναι επιτάπητος, α, μπορεί, μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο. Είναι αδύνατη. Είναι πολιτικά αδύνατον. Οπότε το ερώτημα είναι ποια από τις αδύνατες λύσεις είναι η λιγότερο αδύνατη. Και εγώ θα έλεγα πως η δική μου και όχι μόνο δική μου πρόταση είναι η ε, λιγότερο αδύνατη να εξηγήσω γιατί με δύο τρόπους μπορεί να συμβεί κάτι. Το ένα είναι μια μεγάλη έκρηξη, δηλαδή με κάποιο βαθμό ο βαθμός της κρίσης, η αντίληψη των κινδύνων θα είναι τόσο μεγάλη ώστε θα υπάρξουν πολιτικά κίνητρα και θα γίνει μια επανάσταση αν θέλετε Μία πιθανότητα είναι αυτή και αν γίνει αυτό τότε θα έλεγα πως οι λύσεις ε, τις οποίες υποβάλλω είναι αυτές οι οποίες θα νομοποιηθούν πιο εύκολα ε, ενώπιον των πολιτών. Ευκολότερα θα τις δεχτούν οι πολίτες. Και αυτό μου επιτρέπει να εξηγήσω και κάποια από τα άλλα ζητήματα. Οπότε, κάποιος είπε παραδείγματο χάρη, μίλησε για τους ε, κινδύνους και δυσκολία αποδοχής της αμοιβαιοποίησης του κινδύνου. Αυτό το οποίο εγώ λέω μηχανισμό ε, ασφάλισης, ε, αμοιβαίας ασφάλισης. Αλλά πλέον δεν μιλάμε μόνο για ε, κοινή έκδοση του χρέους, αλλά βασίζεται σε ένα πραγματικό ε, κοινοτικό προπολογισμό με κοινοτικού πόρους που θα βασίζονται σε πλούτο που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορεί να το δεχτούν πιο εύκολα οι πολίτες, γιατί τους λέμε ασφαλίζεις κάτι το οποίο δεν ελέγχεις με μια πολιτική διαδικασία στην οποία δεν συμμετέχεις αλλά πληρώνεις για την ασφάλεια. Λέμε η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει για να διορθώσει τις ασυμμετρίες με τους πόρους που δημιουργούνται από την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Νομίζω πως είναι ευκολότερο αυτό να το δεχτούν οι πολίτες. Ε, αυτές είναι περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να έχουμε ένα γενικό πακέτο. Η εναλλακτική λύση είναι να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κρίση, ότι θα είμαστε επιτυχείς ε, στο να την ε, περιορίζουμε με τις λύσεις αυτές τις εμβαλωματικές. Κάθε φορά δηλαδή δεν πέφτουμε στον κρεμό, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε βαθύτερα αίτια και τις συνέπειες της κρίσης. αν γίνει έτσι δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο να εισαχθούν στρατηγικά κάποια από αυτά τα πέτρα ως ένας μηχανισμός μεταβατικός. Και εδώ πέρα πάλι βλέπω πως ε, αυτό θα μπορούσε να είναι πιο εφικτό να σας δώσω ένα παράδειγμα για την ενισχυμένη συνεργασία και τους ίδιους πόρους και πώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μηχανισμούς για να είναι κάτι πιο πολιτικά εφικτό. Ας υποθέσουμε πως αυτό το συζητάνε οι νομικοί. Το εάν δηλαδή μπορεί να έχουμε ίδιους πόρους και έναν φόρο ε, και ενισχυμένη συνεργασία. Πολλοί νομικοί θα σας πούν πως ε, αυτό δεν γίνεται, η απόφαση για ίδιους πόρους απαιτεί ομοφωνία, πώς μπορεί να συμμετέχουν κάποια κράτη-μέλη με ένα τρόπο στον προπολογισμό και άλλα με άλλο τρόπο. Ας πούμε πώς είναι δυνατόν. Το έχω γράψει, τα έχω γράψει σχετικά στο παρελθόν. Δηλαδή, εάν παραδείγματο χάνει, ας πούμε, τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών και κάποιες χώρες τον επιβάλλουν ε, με ενισχυμένη συνεργασία και συμφωνούν πως θα πάει αυτό για να πληρώσουν τις ε, συνεισφορές τους στον προπολογισμό που υπολογίζονται βάσει του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει πως κάποιες χώρες θα συνεχίσουν να πληρώνουν από τον προπολογισμό τους, άλλες θα συμφωνήσουν ε, σε έναν ε, κοινοτικό φόρο που θα πάει για την συνεισφορά τους. Οπότε δεν θα υπάρξει αλλαγή για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τους ίδιους πόρου. αλλά πολιτικά θα έχουμε φοβερές συνέπειες. Γιατί φανταστείτε πως είστε σε μια χώρα που δεν θα ε, μπει σε αυτό το σύστημα. Οι υπόλοιποι πολίτες δεν πληρώνουν μέσω των προπολογισμών γιατί, γιατί πάει μέσω των φόρων, μέσω του φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Ένα από του λίγου φόρου που θα είναι οι πολίτε και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν να συνεισφέρουν από τον προπολογισμό. Θα είναι δύσκολο μετά για του υπόλοιπου να συνεχίσουν να δικαιολογούν κάτι τέτοιο στου πολίτε του και να λένε Όχι, εμεί πληρώνουμε γιατί δεν θέλουμε να φορολογήσουμε τι τράπεζε. Πολιτικά λοιπόν, αυτό είναι ένα τρόπο όπου μπορεί να εισαχθεί ένα τέτοιο μηχανισμό. Αυτοί είναι δύο τρόποι και, με του δύο τρόπου, είτε όπω είπαμε μια μεγάλη έκρηξη, μια επανάσταση, είτε με μια προσέγγιση πιο σταδιακή νομίζω πως υπάρχει μεγαλύτερη βιωσιμότητα σε κάποιες προτάσεις από αυτές που έκανα σε σχέση με κάποια άλλα πράγματα που ακούστηκαν. Οπότε, επίσης υπάρχουν αρκετά άλλα πράγματα, θα είμαι αρκετά σύντομος. Ε, Παραδείγματος χάρη, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως αυτό είναι ένα ζήτημα ευρύτερο. Εγώ είμαι επικριτικός στο ότι το πρόβλημα της ιδέας είναι η επικοινωνία με τους πολίτες, το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί καμία επικοινωνιακή πολιτική δεν λειτουργεί. Και επίσης, και αλλαγέ στα θεσμικά όργανα είναι πολύ περιορισμένες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επικοινωνεί μέσω των πολιτικών της και της πολιτικής της. Και γι' αυτό εστιάζουμε σε αυτά. Μόνο εάν αλλάξουμε τη φύση της πολιτικής και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει η Ένωση να αποκτήσει μεγαλύτερη ε, και καλύτερη εικόνα στους πολίτες για το τι κάνει και να είναι και πιο υπόλογη γιατί έτσι θα μπορέσει να ε, δώσει στους πολίτες να καταλάβουν το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρόπο σωστό ή και λανθασμένο. Και μία ανησυχία μου ακριβώς σχετίζεται με αυτό το οποίο ανέφερε κάποιο ε, βουλευτής. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε είναι η αντίθετη τάση στο επίπεδο της πολιτικής. Αντί να βλέπουμε μια Ευρω... έναν εξευρωπαϊσμό των εθνικών πολιτικών, έχουμε μια εθνικοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και αυτό με ανησυχεί. Τρία πραγματάκια ακόμα για να προσπαθήσω να απαντήσω έως το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις για το Συμβούλιο και την ε, διαρθρωτική του αμφισημία. Πράγματι είναι δύσκολο να το δούμε αυτό το ζήτημα. Ε, ένα τρόπο βεβαίω είναι μια αλλαγή τη συνθήκης. Μπορούμε να σκεφτούμε να έχουμε παραδείγματο χάρη ένα κοινοβούλιο με δύο σώματα, ένα με ίση εκπροσώπηση των κρατών και ένα με αναλογική. είναι μία από τις άσχημες πτυχές νομίζω της ε, συνθήκης Λισαβόνας είναι η αναλογική εκπροσώπηση στο Συμβούλιο. Οποιοςδήποτε πολιτικός επιστήμονας θα σας πει πως είναι περίεργο να ε, οργανώνουμε αναλογική εκπροσώπηση μέσω τέτοιων μπλοκ. Δηλαδή φανταστείτε πως έχετε μία κοινότητα με τρεις υποκοινότητες μία με 52 άτομα, οι, άλλοι με, οι άλλες δύο με 24 ας πούμε. Και μετά λέμε θα οργανώσουμε την ε, πλειοψηφία, την ψηφοφορία, με συγχωρείτε, αναλογικά με τον πληθυσμό. Δεν έχει το κάθε άτομο μετά η κάθε ψήφος την ίδια αξία, γιατί αυτοί που ψηφίζουν για την κοινότητα των 24 δεν έχουν λόγο. Μόνο αυτοί που ψηφίζουν για την κοινότητα των 52 έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων. Για να σας δώσω ένα ξεκάθαρο παράδειγμα του γιατί ήταν λάθος να οργανωθεί η αναλογικότητα μέσω του ε, μηχανισμού του Συμβουλίου. δεν πολιτικός επιστήμονας ε, το θεωρεί παράλογο. Ε, αυτό ίσως είναι κάτι που πρέπει να ξανασκεφτείτε και ίσως είναι ένα κίνητρο για να κάνετε μία αλλαγή της συνθήκης. Αν δεν υπάρχει αλλαγή της συνθήκης, η άλλη λύση είναι, όπως είπα, μέσω μεγαλύτερου πολιτικού κεφαλαίου στην Κομισιόν με το να συνδεθεί δηλαδή με τις ευρωεκλογέ. Μόνο έτσι το, το βλέπω εγώ. Τελευταίες δύο ερωτήσεις. Για το εάν θα ήταν αποτελεσματικό να μετατραπούν οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν εκλογική αναμέτρηση για τον πρόεδρο της Επιτροπής. Εδώ ίσως τα εθνικά πολιτικά κόμματα να συνεχίσουν να ελέγχουν τις εκλογές αυτές επί τη βάση εθνικών πολιτικών θεμάτων. Η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ εμπειρική βέβαια. Οι δικές μου προσδοκίες είναι ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Αν συμβεί, γιατί να μην δοκιμάσουμε αυτό το οποίο προτείνω. Αν ο κόσμος μπορεί να προχωρήσει σε ελεκτικές εκλογικές διαδικασίες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο, γιατί να μην το κάνει. Ο λαός σας αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ενδιαφερθεί για τα κοινοτικά. Ένα τελευταίο σημείο για τις κοινέ ταυτότητες που θα πρέπει να προηγηθούν και όχι να ακολουθήσουν την δημιουργία των πολιτικών κοινοτήτων. Ο Χόμπς σε σχέση με τις πολιτικές κοινότητες είχε πει ότι οι κοινότητες αυτές είναι κάτι το οποίο δημιουργείται από το εσωτερικό των συγκρούσεων των γειτόνων. Σαν συνέπεια πιθανών συγκρούσεων λόγω της κατανομής του κοινού χώρου να προχωρήσει σε συνεργασίες. Αυτό έχει άμεση σχέση βέβαια και με την προηγούμενη ύπαρξη μιας πολιτικής ταυτότητας και έχει άμεση επίσης σχέση με τον τρόπο αντιμετώπισης της σύγκρουσης και του προβλήματος. Το ερώτημά μου είναι, εάν η αλλολοεξάρτηση περάσει σε διαφορετικό επίπεδο, τότε οι πολιτικές κοινότητες πρέπει να ακολουθήσουν. Αν δεν γίνει αυτό, τότε χειροτερεύει το θέμα της ε, ε, αντιπροσώπευσης της δημοκρατικής. Οι ταυτότητες, οι ιστορικές, οι πολιτικές είναι κοινωνιολογικές προϋποθέσεις οι οποίες ευνοούν την λειτουργία, την εύρυθμη της πολιτικής κοινότητας. Αλλά η ανάγκη για μια πολιτική κοινότητα γεννιέται από την αλληλοεξάρτηση, από την κοινωνική σύγκρουση και από τις αμοιβαίε μορφές εξωτερικής αντιπροσώπευσης που δημιουργεί ο πολίτης όταν μοιράζεται ένα συγκεκριμένο χώρο πολιτικό ή οικονομικό. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε εδώ είναι να κατανοήσουμε ότι μοιραζόμαστε έναν ενιαίο χώρο, κοινό χώρο και θα πρέπει εμείς να ασκήσουμε τη διακυβέρνηση του συγκεκριμένου αυτού χώρου τις εξωτερικότητες αν θέλετε προς το κοινό συμφέρον. Ευχαριστώ λοιπόν όλο τον κόσμο και ευχαριστώ και τους διευμηνείς που έμειναν περισσότερο από ό,τι συνήθως. Ευχαριστώ και καλές διακοπές. Αυτή ήταν η τελευταία συνεδρίασή μας πριν το Σεπτέμβριο.